Καλώ Καλώς ήρθατε όλοι στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Παρακαλώ λοιπόν να σταματήσετε τις συζητήσεις και να καθίσετε διότι έχουμε αρκετά γεμάτο πρόγραμμα. Πρώτο θέμα στην απογευματινή ημερήσια διάταξη είναι το σημείο υπαριθμών 11 εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Και δίνω κατευθείαν τον λόγο στον εισηγητή μας, τον Ταμιάνο Ζοφόλη. Παρακαλώ. Ταμιάνο, μ' ακού? Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή αποτελεί μια απάντηση του Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική χαμηλής κυνηγικότητας. Συναρμόδιες οι ΤΡΑΝ και οι ΕΜΒ επιτροπέ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του κανονισμού. Η βιώσιμη λοιπόν κινητικότητα αποτελεί ένα από τα κυριότερα στοιχεία μια ευρύτερη μετάβαση προ ένα μοντέλο ανάπτυξη που αναζητάμε ως Ευρωπαίοι στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας με εκπομπές άνθρακα αντίστοιχε ώστε να παραμένει η ανταγωνιστική ένωση, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και για να τηρηθούν οι ανάγκες κινητικότητας ατόμων και αγαθών. Η πρόκληση λοιπόν αυτή συνίσταται στο να καθορίσουμε και να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα νέα μέτρα για την ανάπτυξη μεταφορών που θα τροφοδοτούνται από εναλλακτικέ μορφές ενέργεια με χαμηλέ εκπομπε τρύπων, τοπικά και σφαιρικά. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι σήμερα συμβάλλουν στο στο τέταρτο της εκπομπε ρήπων θερμοκηπίου και αποτελούν, οπω ξέρουμε, την κύρια πηγή ατμοσφαιρικής δρύπανσης. Ο στόχος που είχαμε είναι ξεκάθαρος. Μέχρι το 2050 οι εκπομπές θερμοκηπίου από τις μεταφορές θα πρέπει να είναι κάτω από το 60% σε σχέση με το 1990 και διαδοχικά θα πρέπει να προσεγγίσουν το 0. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα θέμα πολύ λεπτό και ευαίσθητο που θέλησα να προσεγγίσω με λίγες σειρές περιλαμβάνοντας κάποιες θεματικές που συζητούνται εδώ αλλά και σε άλλες επιτροπές όπως η νέα οδηγία για τις ΑΠΕ όσον αφορά τα βιοκαύσιμα κανονισμός για την ταξινόμηση και παρακολούθηση των οχημάτων που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στην Ολομέλεια. Έχω πρόθεση να συντονιστώ και με τους άλλους συναδέλφους, ώστε να βρούμε συγκεκριμένες και απτές λύσεις. Η γνωμοδότης προσεγγίζει το θέμα των εκπομπών σε σχέση με διάφορα οχήματα. Φορτηγά, αλαφρά οχήματα, αυτοκίνητα, γεωταχή. πολύ συνθετικά, πολύ σύντομα. Και προτείνω τα εξής να θέσουμε στόχο εκπομπών δεξιδίου άνθρακα για τα αυτοκίνητα μεταξύ 68 και 78 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο για τα μικρά φορτηγά 120. 100-120. Όπως εξάλλου ήδη έχει ζητηθεί δηλαδή παλαιότερα από το Κοινοβούλιο. Επίσης ζητάμε να αναπτύξουμε το ταχύτερο δυνατό ένα τεστ οδικό το οποίο θα είναι ρεαλιστικό και διαφανές ώστε να υπάρχει ένας θαραλέο στόχος για να ενθαρρύνουμε την είσοδο στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με τη χρήση μπαταρίας δεύτερης γενιάς. Επίσης, είναι απαραίτητο να εργαστούμε πάνω σε ένα σύστημα σήμανσης περισσότερο διαφανές όσον αφορά την κατανάλωση των καυσίμων. Όσον αφορά τώρα τα βαρέα οχήματα, και εδώ υπάρχει ένα κενό πολύ σημαντικό, ζήσα από την Κομισιόν να εκπονήσει μια πρόταση σε σχέση με την παρακολούθηση των εκπομπών στα βαρέα, οχή, στα οχήματα μέχρι το τέλος του τρέχοντο έτους, το 2017, και να προταθούν στόχοι φιλόδοξοι εκπομπών διοξιδίου. Να τονίσω εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες οχημάτων ξεκάθαρα όρια όσον αφορά τις εκπομπές. Παρόλο που εκπροσωπούν βεβαίως περίπου το 1 τέταρτο εκπομπών διοξιδίου άνθρακα που προέρχεται από τι μεταφορές. Σε σχέση τώρα με τις ταξινομήσεις, σύμφωνα με τι υπάρχουσες συζητήσει, ξαναπροτείνω ένα σύστημα ταξινόμησης περισσότερο διαφανές, το οποίο θα περιλαμβάνει βεβαίως και την ε, εποπτεία ώστε να καλύψουμε και τα κενά που ανέκυψαν με το Dieselgate. Για την αεροπλοεία εξέφρασα τις αμφιβολίες σε σχέση με τους χαμηλούς στόχους του περασμένου φθινοπόρου στα πλαίσια της ΕΚΑΟ, ιδιαίτερα όσον αφορά τους στόχους για το διοξίδιο που θα ισχύσουν το 2020 και μετά και κυρίως για το εθελοντικό τους χαρακτήρα από το 2021 μέχρι το 2026. Και έχουμε και τη νέα πρόταση της ε, Κομισιόν που για, τους, για τις πτήσεις της εσωτερικής της Ένωσης έχει ακολουθήσει ένα σύστημα διαφορετικό. Παρόλο που ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί το μόνο δρόμο, το μόνο υπαρκτό δρόμο για μια πιο φιλόδοξη στοχοθέτηση. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το υπάρχον τωρινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για να μειώσουμε τι αγκομπές του άνθρακα. Μετά, για τι θαλάσσιε μεταφορέ, περίλαβα αυτό που ήδη έχει κάνει το Κοινοβούλιο για τις μεταφορές Θεωρώ ότι εδώ δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών ρήπων θερμοκηπίου και αυτό ακριβώς το λόγο θα είναι απαραίτητο ελήψη συγκρίσιμων μεθόδων διεθνώς, οι εκπομπές ε, διοξιδίου στα λιμάνια της Ένωσης από και προς τους λιμένες αυτούς, θα πρέπει λοιπόν να μπουν αυτοί οι ρήποι στο σύστημα TS από το 2023 και μετά. Όσον αφορά τώρα την υπέρβαση των ε, καυσίμων πρώτη γενιάς Ζήτησα πιο αυστηρού στόχου σε σχέση με αυτού που προβλέπονται στη νέα οδηγία για τι ανανεώσιμε, που θα λαμβάνουν υπόψη του τι αλλαγές κατεύθυνση όσον αφορά την χρήση διασφαλίζοντα βεβαίω την ε, προστασία των επενδύσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Επίσης ζητώ μια ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά των πιο προηγμένων βιοκαυσίμων που όμως θα πρέπει να ακολουθούν την ιεραρχία των απορριμμάτων και θα πρέπει να τηρούν βεβαίως ισχυρά κριτήρια βιωσιμότητας ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα τα οποία είχαμε στο παρελθόν με τα καύσιμα της πρώτης γενιάς. Τέλος, και εδώ καταλήγω, υπογραμμίζω το ρόλο του αερίου στην μετάβαση προς την αποανθρακοποίηση των μεταφορών και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι έχω πρόθεση να καταθέσω κάποιες πληρωματικέ τροπολογίες για το κείμενο για να απτύξουμε καλύτερα κάποια στοιχεία και να περιλάβουμε νέα που για λόγους έλλειψης χώρου δεν μπόρεσα να περιλάβω. Ενημερώνω τους ε, συναδέλφους ότι 3η Μαΐου είναι η προθεσμία της τροπολογίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ζόφολη, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Το τελευταίο 12 ε, ασχοληθήκαμε πολύ με τις εκπομπές, ε, μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή ΕΜΙΣ, όπου έχουμε εντοπίσει τέσσερα θέματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς. Ε, διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι μετρήσεις σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τις εκπομπές όχι μόνο στο εργαστήριο. Νομίζω ότι σίγουρα θα είναι χρήσιμη εδώ η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ε, θα μπορέσουμε έτσι να ρυθμίσουμε τις εκπομπές ε, του αζότου, οξυδίων του αζότου. Όταν μιλάμε εδώ για μείωση των εκπομπών θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ντίζελ αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Ε, κύριε Τσόφολη, ε, εδώ γνωμοδοτούμε ενώ ε, ε, ε, επί της, αρμο... επί αρμόδια είναι η Επιτροπή Μεταφορών. Θέλουμε λοιπόν μια ισορροπημένη έκθεση. Έχουμε μια ενιαία στρατηγική στην Ευρώπη και λέμε ότι πρέπει να προβλέπετε συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ για την ε, βιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στη βιομηχανία και το περιβάλλον. Ο συνάδελφος Έικχοτ είναι παρόν. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλά στοιχεία στην ε, πρόταση που εμένα μου δημιουργούν προβλήματα. Μιλάμε για την απαλωτρίωση, όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών. Ε, μας ενδιαφέρει το μέλλον των μεταφορών. Πρέπει εμείς ως βουλευτές να το αποφασίσουν αυτό ή θα πρέπει να αφήσουμε την αγορά να αποφασίσει, δηλαδή να διατεθούν ε, τα προϊόντα στην αγορά και ο καταναλωτής ε, να αποφασίσει. Ως πολιτικοί θα πρέπει εμείς να ορίσουμε το πλαίσιο για καινοτόμα και βιώσιμη πολιτική δεν ε, νομίζω ότι η ε, ενιαία οικονομία θα αποτελέσει ε, εδώ την κατάλληλη λύση. Να λέμε το να υποδεικνύουμε συγκεκριμένο ποσοστό σε ποια βάση βασίζεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και τις απαραίτητες υποδομές, για παράδειγμα, αν θέλουμε συγκεκριμένο ποσοστό ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε εμείς ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο και για τις καινοτομίες. Όσον αφορά τις ε, αερομεταφορές, ο κύριος Ζόχολη αναφέρθηκε εν μέρη στο θέμα αυτό. Οι προτάσεις της ε, Επιτροπής Μεταφορών είναι πολύ πιο ευρείες. Στις αερομεταφορές έχουμε διεθνή ανταγωνισμό και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούμε και στις συνθήκες πλαίσιο, τουλάχιστον να μην τις αγνοούμε. Αγαπητέ συνάδελφε, αναφερθήκατε στα 68 γραμμάρια. θέλουμε να, έχουμε τις, να χρησιμοποιούμε τις νέες παγκοσμίως νορμασμένες διαδικασίες δοκιμών για τα ελαφρά οχήματα, WLTP. Ε, ίσως λοιπόν δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με ε, συγκεκριμένα όρια, αλλά να ορίσουμε ποσοστό, κάτι που είναι πολύ πιο ρεαλιστικό. Όσον αφορά τις ε, υποχρεωτικές ρυθμίσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να υποδείξουμε τους ε, στόχους, ε, αλλά εάν επιμείνουμε σε δεσμευτικούς στόχους, ε, μέχρι το 2030 δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να τους πετύχουμε. Τέλος, όσον αφορά την ηλεκτροκινητικότητα, δεν αποτελεί πανάκια, διότι από πού προέρχεται το ρεύμα. Εάν θέλουμε ε, κατά 25% ε, ηλεκτροκίνητα οχήματα. Εάν το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται ε, από λιγνίτη, για παράδειγμα, τότε δεν είναι βιώσιμη η ενέργεια αυτό το πράγμα. Στην κάτω Σαξονία η Audi έχει μια καινοτόμα προσέγγιση. Από το πλεόνασμα αιωλικής ε, και ηλιακής ε, ενέργειας ε, παράγουν μεθάνιο για την ηλεκτρική κίνηση των οχημάτων. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες προς διάφορες κατευθύνσεις και τελικά ο καταναλωτής θα μπορεί έτσι να επιλέξει το πιο βιώσιμο προϊόν. Προσλέπω στη συζήτηση με τους συναδέλφους. Νομίζω ότι θα είναι πολύ επικοδομητική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τέμες Μάκερ από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Σοφόλη. Συνάδελφοι, βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των μεταφορών στις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Το επιβεβαίωσε και η υπηρεσία περιβάλλοντος και ειδικά οι οδικές μεταφορές παίζουν μεγάλο ρόλο και είναι μία από τις κύριες αιτίες Τη ρήπανση του αέρα στις ε, πόλεις μας, η οποία ρήπανση σκοτώνει και βλάπτει και το κλίμα και τον άνθρωπο και την οικονομία. Είναι τεράστια η επίδραση της αρνητική και Βεβαίω έχουμε τι ιδιαίτερα ευπαθεί ομάδε. Πάνω από 400.000 πολίτε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρουν κάθε χρόνο από την άσχημη ποιότητα του αέρα. Τώρα, για την μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και κοινωνία, θα πρέπει να δούμε το τι θα κάνουμε στον τομέα της ε, κινητικότητας. Πρέπει να σκεφτούμε κάποιες εναλλακτικές, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και βεβαίως να τα πλαισιώσουμε αυτά. Καλώς ορίζω οπωσδήποτε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περιέχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Η Κομισιόν σωστά τονίζει ότι ε, αυτό παρουσιάζει και πολλές ευκαιρίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σοφόλη. Δεν είναι εύκολα αυτά τα οποία έκανε και βεβαίω είναι πολύ εκτεταμένο και το πεδίο εφαρμογής και θα ήθελα να εγώ να συνεισφέρω όσο μπορώ στην υποδομητική αυτή η έκθεση. Θα πρέπει, όπως είπαμε, να τονιστεί περισσότερο το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σύνεπείς με τις συστάσεις της, της Διερευνητικής Επιτροπής ΕΜΙΣ ε, την έκθεση της οποίας ενέκρινε και η Ολομέλεια. Εκεί πέρα περιέχουν κάποιες, περιέχονται κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις για το πρασίνισμα των μεταφορών, για μια προδιαγραφή Euro 7, για το πώς γίνονται οι δοκιμές έγκρισης τύπου και για το θέμα των καταναλωτών και βέβαια με την απαραίτητη σύνδεση με την κυκλική οικονομία Και βεβαίως αυτό για μένα περιέχει το θέμα της ε, μετάβασης και της αυθόρμητης μετάβασης ε, προς μια διαφορετική κινητικότητα και βεβαίως να δούμε και την διατροπική κινητικότητα με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Θα καταθέσω λοιπόν και κάποιες ε, τροπολογίες και αναμένω μια γρήγορη και καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την άλλη τον λόγο έχει τώρα η κυρία Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης που καλύπτει τα βασικά θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει ή θα ξεκινήσουμε προσεχώς να συζητάμε. Θα αναφέρω π.χ. τα όρια εκπομπών, τις μετρήσεις γιοταχή και φορτηγών, εγκρίσει τύπου, τη συμπερίληψη αεροπορίας και ναυτιλίας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως καύσιμα και αν και πρέπει να συζητήσουμε ακόμα κάποιες προτάσεις. Το σχέδιο αυτό θέτει τις βάσεις έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να εκφράσει τουλάχιστον τις προσδοκίες του. Αφενός, θα ήθελα να θέσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Στην παράγραφο 14 ο εισηγητής ζητάει πρώτα απ' όλα αύξηση των ανωτάτων τιμών για το βιοκαύσιμα της, ε, σε σχέση με τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς. Θα ήθελα να πω πως ε, τα οικοπροϊόντα που προκύπτουν εδώ πέρα περιέχουν και σημαντικές ε, πρωτεΐνες για τις ζωοτροφές. Στην παράγραφο 15 ο εισηγητής, την οποία χαιρετίζω, ζητάει από την Κομισιόν να προστατεύσει τις υφιστάμενες επενδύσεις στα δύο καύσιμα. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ λοιπόν υπάρχει μια αντίφαση. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας εξηγήσει τις δύο παραγράφους αυτές, ανεξαρτήτως του ότι δεν θέλω να μπω στις ε, λεπτομέρειες. Απλά να δούμε τη γενική εικόνα. Ο κλάδος των μεταφορών ευθύνεται για 25% των εκπομπών και εξακολουθεί να εξαρτάται κατά 94% από ορυκτά καύσιμα και είναι ο μοναδικός κλάδος στον οποίο οι εκπομπές τα τελευταία 25 χρόνια αυξήθηκαν. Τσέτερης πάρυμπους ε, βλέπουμε ότι πάλι καμία αλλαγή δεν θα υπάρχει γιατί από ό,τι φαίνεται τις επόμενες δεκαετίες η μεταφορά και ανθρώπων και εμπορευμάτων θα αυξηθεί. Έχουμε λοιπόν μεγάλες φιλοδοξίες, θέλουμε η κοινωνία μας μέχρι τα μέσα του αιώνα να έχει απαντρακωθεί και ελπίζουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Και στη συζήτηση για το πώς ε, θα χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως κάψιμα, ακούω γιατί αυτό και όχι το άλλο, δεν είναι καλή λύση, ή μιλάμε για ποσότητες ομοιοπαθητικής, ελάχιστα ποσοστά. Τουλάχιστον ε, για την χρήση ηλεκτρισμού όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές, είναι τελείως μη ικανοποιητικέ οι προτάσεις εδώ πέρα. Πρέπει λοιπόν να μην σκεφτόμαστε ότι υπάρχει μία λύση η οποία θα ε, λύσει όλα τα προβλήματα. Ακούγοντας αυτές τις συζητήσεις έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή στο θέμα της ε, κινητικότητας ε, του μέλλοντος χανόμαστε σε μικρά βήματα χωρίς να ξέρουμε πού μας οδηγεί το ένα βήμα μετά το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι οι δυνατότητες αυτής της έκθεσης δεν είναι στο να αποφασίσουμε από τώρα ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες των επόμενων 15 ετών. Είναι το να δούμε ακριβώς τη γενική εικόνα. Πού είμαστε, πού θέλουμε να είμαστε σε μερικές δεκαετίες και ποιες συστημικές αλλαγές πρέπει να επιφέρουμε. Λοιπόν. οι σωστές άλλαγες της ε, πορείας θα ωφελήσουν μόνο αν ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Γι' αυτό ελπίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, αντί για ποσοστά και στόχους ε, σε δεκαδικά ψηφία. Χαίρομαι λοιπόν, αναμένω την συνεργασία. Θεωρώ ότι Υπάρχει αρκετή καινοτομία στη βιομηχανία και χρειάζεται χρόνος βεβαίως για να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη τα οποία θα μας οδηγήσουν στο μεγάλο στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σκιώση, συγγήτρια της ΓΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Τζοφόλη, για αυτό το σχέδιο έκθεσης όπου αναφέρεται σε διάφορους τρόπους ε, μεταφορών. Θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ε, και αναφέρεται ιδιαίτερα στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Αυτή τη στιγμή η πολιτική μεταφορών στην Ευρώπη στηρίζεται κυρίως στην ε, μείωση των εκπομπών ε, με τη χρήση νέων τεχνολογιών όσον αφορά τα καύσιμα και τα οχήματα. Τα τελευταία χρόνια όμως ε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στην βιομηχανία αυτοκινήτων που οδήγησαν σε αμφισβήτηση της ε, δέσμευσης, ε, της αφοσίωσης ε, της βιομηχανίας αυτοκινήτων να μειώσει τις εκπομπές. Νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να μειώσουμε τις εκπομπές όχι μόνο με χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και με άλλους τρόπους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πετύχουμε τους στόχους μας είναι η εφαρμογή ε, ε, μιας ευρείας δέσμης μέτρων που να συμπεριλαμβάνει την σωστή χρήση γης, ε, το να πηγαίνει κανείς με τα πόδια ή να παίρνει το ποδήλατο. Πολιτικές που μπορούν να συμπληρώσουν και να στηρίξουν τις νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες ε, που μας παρέχονται με τα ψηφιακά μέτρα και γνωρίζοντας ότι και οι τιμές παίζουν ρόλο κατά την επιλογή μέσου μεταφοράς. Η κινητικότητα όπως διαμορφώνεται στις μέρες μας συνδέεται με τη χαμηλή τιμή του πετρελαίου. Αυτός ο παράγοντας ε, έχει επιβραδύνει την μεταφορά σε τρόπο ε, μεταφοράς ε, ε, χαμηλών εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διάφορα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπουν τη διάθεση σημαντικών χρηματικών ποσών και νομίζω ότι είναι απαραίτητο τα διάφορα προγράμματα και τα διάφορα μέσα να εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότησης για προγράμματα που συνδέονται με τη μεταφορά για την μετάβαση σε τεχνολογίες χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η μείωση των εκπομπών στις μεταφορές ε, είναι θέμα που εναπόκειται στις εθνικές ε, και ακόμα και σε τοπικές αρχές. Σε αστικές περιοχές το 23% των εκπομπών στην Ευρώπη προέρχονται από αστικές μεταφορές. Η προβληματική αστική πολιτική λοιπόν είναι ένας παράγοντας όπου όμως δεν έχει καμία επιρροή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ισχυρό συντονιστικό ρόλο για να μπορέσει να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των αστικών μεταφορών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και η ψηφιοποίηση έχουν καταστήσει δυνατούς νέους τρόπους κινητικότητας που μπορεί να καταστήσουν λιγότερο απαραίτητο ή χρήσιμο το να έχει κανείς στην κυριότητά του αυτοκίνητο. Θα ήθελα να δοθεί περισσότερη ορατότητα στις νέες λύσεις για την κινητικότητα εντός και μεταξύ πόλεων. Το κόστος επίσης των νέων τρόπων μεταφοράς θα πρέπει να είναι πιο διαφανές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο είναι ένα χρήσιμο καύσιμο για την περίοδο μετάβασης, μόνο όμως ως τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τα τερματικά υποδομή που δημιουργείται για το υγροποιημένο φυσικό αέριο να μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για βιοκαύσιμα. Δεν νομίζω ότι αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Θα το συμπεριλάβω όμως σε δική μου τροπολογία. Προσλέπω στην καλή συνεργασία με τους συναδέλφους πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι ένα θέμα που με παθιάζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Keith Taylor ε, θα μιλήσει για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζωφόλη για το σχέδιο γνωμοδότησής του και να τον συγχαρώ που προτείνει κάποιες πολύ χρήσιμες προσεγγίσεις. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επικροτήσω την έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για στόχο μείωσης ε, του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2020 για ελαφρά οχήματα. Με βάση τις δοκιμές ε, υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης ε, και όλα αυτά προς όφελος των καταναλωτών. Ε, θα παρακαλούσα να μιλάτε πιο σιγά, διότι ε, δεν ακούγομαι. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες που ελπίζω ότι θα βελτιώσουν την έκθεση αυτή. Ο τομέας μεταφορών στην Ευρώπη είναι ο μόνος που δεν έχει καταφέρει να μειώσει τις κλιματικές επιπτώσεις του την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 27% από το 1990 και οι μεταφορές αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 13% των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορέσουμε λοιπόν ε, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την ε, Συμφωνία του Παρισιού θα πρέπει να μηδενιστούν μέχρι τα μέσα του αιώνα. Επίσης ο τομέας αυτός ε, αντιπροσωπεύει το 70% της κατανάλωσης πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως ε, λόγω της ραγδαίας αύξησης των οδικών μεταφορών και αερομεταφορών. Είναι σαφές ότι ο τομέας μεταφορών της Ευρώπης βρίσκεται σε μη βιώσιμο δρόμο που διακυβεύει έτσι το κλίμα, την υγεία μας και την ποιότητα ζωής μας. Εάν δεν αλλάξουμε τα πράγματα στον τομέα της κινητικότητας, ε, θα αυξήσουμε την εξάρτηση της Ευρώπης από το εισαγόμενο πετρέλαιο και ε, θα ε, υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε στο μέλλον ενεργειακή κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να εσωτερικεύσουμε το εξωτερικό κόστος των μεταφορών. Για παράδειγμα, η, ε, ε, ε κυροζήνη για τα αεροπλάνα ε, που είναι αφορολόγητη, αυτό είναι μη δίκαιος ανταγωνισμός, είναι δηλαδή ένα άδικο πλεονέκτημα υπέρ του τομέα μεταφορών. Επίσης, η ατμοσφαιρική ρήπανση που συνδέεται με ασθένειες καρδιαγγειακές και αναπνευστικές οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταφορές. Και καταλαβαίνω ότι η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στην μείωση των εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα, αλλά δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τις ε, σημαντικές ανθικές επιπτώσεις της ρήπανσης του αέρα η κακή ποιότητα του αέρα που, που αναπνέουμε είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις αστικές περιοχές και η αυξημένη χρήση του ντίζελ αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για την υψηλή συγκέντρωση σωματιδίων στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπιστώνει ότι το ντίζελ είναι καρκινογενή ουσία. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε τη δυνατότητα απαγόρευσης διζελοκινητήρων. Διότι όχι μόνο επιδεινώνεται έτσι η ποιότητα του αέρα, αλλά ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και μόνο από το 2013 μέχρι το 2030 προβλέπεται ότι το κόστος ε, θα είναι 307 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το 80% των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύντομα θα ζουν σε αστικές περιοχές ε, και η αστική κινητικότητα αντιπροσωπεύει το 70% των ρήτων και το 40% προέρχεται από τις οδικές μεταφορές και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό δείχνει πόσο απαραίτητο είναι να κινηθούμε προς πιο βιώσιμες ε, μορφές μεταφορών. Και να πω και κάτι πιο θετικό, είμαι πεπισμένος ότι αυτά τα συστήματα αστικών μεταφορών ε, θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών. Το 60 τα 100 των ε, ε, ε, μεταφορών εντός των πόλεων είναι λιγότερο από 6 χιλιόμετρα και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε μη μηχανοκίνητους τρόπους μεταφορών, όπως είναι το να πηγαίνει κανείς με τα πόδια ή το να παίρνει το ποδήλατο. Επίση, ω συνεπιβατισμό και να έχουμε και βιώσιμες μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς. Ε, αυτοί είναι τρόποι να έχουμε μια βιώσιμη αλυσίδα μεταφορών. Η υπερβολική εξάρτηση της, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης από τις οδικές μεταφορές είναι επίσης ένα πρόβλημα. Η βελτιωμένη εφοδιαστική, ιδιαίτερα όσον αφορά τις, τον την τελευταία αλυσίδα στις ε, μεταφορές ε, θα βελτιώσει σαφώς την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε λύση για τα σημεία συμφόρησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για βελτίωση εδώ. Μπορούμε να μειώσουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τους επικίνδυνους ρήπους στον αέρα που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τους συναδέλφους για να πετύχουμε μια καλή λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύη για το EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον Σένφο Τζόφολη για την ομοδότησή του. Πρώτη γενική παρατήρηση θα ήθελα να κάνω αναφέρθηκε και από τους άλλους συναδελφούς. Αυξάνονται εκπομπές λοιπόν στον τομέα των μεταφορών και έχουμε πολλά στοιχεία και εκθέσεις που το αναφέρουν. μεταξύ αυτών και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Είχαμε και το θέμα της απάτης των διαφόρων κατηγοριών με το Dieselgate που εξετάσαμε για ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο. Δέχομαι με μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά την έναρξη διαδικασία σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα και τους ρήπους, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Συμμερίζουμε επίσης και το αίτημα για βελτίωση όλου του συστήματος ελέγχου και συμμόρφωση των χυμάτων στον δρόμο. Να μην δούμε δηλαδή μόνο κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση, αλλά να μειώσουμε τους δελεστές συμμόρφωσης στο χαμηλότερο δυνατό αριθμό, γιατί ο συντελεστή ε, συμμόρφωση θυμάμαι ότι ήταν μια πολιτική απόφαση που λήφθηκε για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα. Σε πλήρη αντίθεση δηλαδή με τα δεδομένα τα υπαρκτά των τεχνολογιών σήμερα που επιτρέπουν ακριβώς να περιοριστούν τα όρια. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να εξετάσουμε περισσότερο στο Κοινοβούλιο εδώ την αρχή της επιστημονική ουδετερότητας στην οποία είμαστε προσκολλημένοι και που μας οδήγησε σε λάθος δρόμο. Είναι αδιανόητο σήμερα να θέλει κανείς να ακολουθήσει την αρχή αυτή και να μην καταλάβει ότι είναι απαραίτητο να προωθήσει τις πιο καθαρές τεχνολογίες με χαμηλότερο αντίκτυπο τα φίλτρα ας πούμε σε σχέση με τους κινητήρες diesel. Και η Κομισιόν, αναρωτιέμαι, έχει πρόθεση να διερευνήσει αυτό το θέμα για το οποίο υπάρχει ακόμα μεγάλη σύγχυση. Και τη στιγμή μάλιστα που έχουμε σήμερα δεδομένα που μας αποδεικνύουν ότι δεν φιλτράρονται ακριβώς αυτά τα σωματίδια, απλά και μόνο διασπώνται σε μικρότερα σωματίδια, κάτι το οποίο προκαλεί βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Δεν μιλάμε και για την ηχητική ρήπανση. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό, που προκαλεί νεκρούς και θύματα κάθε χρόνο. Κάτι για το οποίο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αντίθετα, να πω ότι δεν συμφωνώ με τον εισηγητή όσον αφορά την ένταξη του σήματος στίες για, το, για τις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει να δούμε αν ανατομέα, θαλάσσιες μεταφορές ή αεροπλοεία, αν θα μπορέσουν να υπάρξουν πιο συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Ένα απλό παράδειγμα εδώ για τις αερομεταφορές είναι το ότι έχουν αυξηθεί οι εκπομπές χωρίς καμία ουσιαστική βελτίωση. Και το κόστος το πληρώνουν οι καταναλωτές, όσοι δηλαδή από μας αγοράζουν το ειστήριο. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε ακριβώς αυτές τις ποσοστώσεις. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες δράσεις βέβαια, ιδιαίτερα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, τομέας που έχει μείνει πολύ πίσω και που παρουσιάζει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και φορολογική μόχλευση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρήση κινητήρων με καύσιμα που ρηπαίνουν λιγότερο όπως το φυσικό αέριο. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες μεταφορές ακόμα και τα πανιά, παλιός τρόπος μεταφορών αυτών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σήμερα ακόμα. Πάντως, με χαρά διάβασα στην ανακοίνωση της Κομισιόν ότι λέει επιτέλους της Κομισιόν ξεκάθαρα ότι είναι απαραίτητο και καλεί τις χώρες μέλη να εξαλείψουν τις άμεσες και έμεσες ενισχύσεις στα ορυκτά καύσιμα. Γιατί υπάρχουν χώρες μεταξύ αυτών και η Ιταλία που συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να αξιοποιηθεί και ο σιδηρόδρομος αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτά βλέπω εγώ ως τελικά συμπέρασμα αυτή την ομάδα Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. κυρία Ντορνάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ζόφελ για τη δουλειά του. Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες. Συγκεκριμένα είμαι υπέρ Στοχοθέτηση για μετά το 2025 για τα οχήματα και τα μικρά φορτηγά νέου κύκλου, ώστε να εναρμονιστούμε με τα παγκόσμια ισχύοντα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τονίσω για αυστηρότερη συμμόρφωση, όπως ακριβώς μας είπαν δηλαδή οι εμπειρογνώμονες του Παγκοσμίου Φόρουμ, όσον αφορά τα οχήματα. Όπως είπε εξάλλου και ο ΙΕ σε σχέση τώρα με την θέσπιση ενός νέου κύκλου δοκιμών, θα πρέπει να, να προσέξουμε εδώ την αμοιβαιότητα εφαρμογής αυτού του νέου κύκλου δοκιμών παγκοσμίω στις ασιατικές χώρες και στην Αμερική συγκεκριμένα. Συμφωνώ βεβαίω για την πρωτοβουλία όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες νέας γενιάς. Θα πρέπει, μαζί με τις χώρες που το επιθυμούν, να συντονιστούμε και να δράσουμε, όχι μόνο στην Ένωση, γιατί οι διεθνείς ε, προδιαγραφές εδώ είναι απαραίτητες. Τώρα, όσον αφορά τη διαφάνεια στις, ε, στη σήμανση, θα πρέπει να υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα για τους καταναλωτές όσον αφορά τα, τις εκπομπές και τα καύσιμα και θεωρώ ότι εδώ και πάλι θα μπορούσαμε να βοηθηθούμε από τους διεθνείς οργανισμούς. Τώρα για την εποπτεία και την παρακολούθηση σχετικά με τα βαρέα οχήματα και την μείωση των εκπομπών για την περίοδο μετά το 2025, θεωρώ ότι η Κομισιόν και πάλι θα πρέπει να στηρίξει δράσεις στα πλαίσια του Παγκοσμίου Φόρου που ανέφερα προηγουμένω. Όσον αφορά τα αστικά λεωφορεία με χαμηλές εκπομπές δρύπων θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ώστε να διευκολύνουμε την εφαρμογή οικολογικών κριτηρίων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Μετά το Dieselgate θα πρέπει επίσης να εποπτεύουμε πιο αυστηρά την αγορά, ιδιαίτερα για τα σωματίδια και όπως λέει και το Παγκόσμιο Φόρουμ να προχωρήσουμε προς μια εναρμόνιση των προδιαγραφών για αυτά τα αρχήματα... Θα πρέπει λοιπόν μετά από αυτό το σκάνδαλο να υπάρχει μια αναμασμένη προσέγγιση. Τώρα για του παράγοντε συμμόρφωση, για το άζωτο και τι εκπομπέ αζώτου που θεωρούνται υψηλέ θα πρέπει να επανεξεταστούν, αλλά μόνο στο μέτρο όπου η εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων ισχύει και σε άλλες περιοχές κόσμου, ιδιαίτερα στι περιοχέ όπου υπάρχει αυτοκινητοβιομηχανία που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κλιματικούς στόχους για το 2030 και στόχους που θα απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού στα πλαίσια της διεθνούς αεροπλοείας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τις ε, θέσεις του Διεθνού Οργανισμού ε, για τη θάλασσα όσον αφορά τις εκπομπές και θα μπορούσαμε εκεί να ενθαρρύνουμε ακριβώς τα μέτρα τα οποία απολέπουν στη μείωση της εκπομπής ρήπων στους διεθνείς λιμένες. Ο στόχος μας βέβαια παραμένει το να να πετύχουμε την απαθρακοποίηση του... στον τομέα των μεταφορών, αλλά όλα αυτά δεν θα γίνουν χωρίς συντονισμό μεταξύ κρατών στα πλαίσια δομών διεθνών που θα είναι ε, νόμιμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις. Λόγω λήψης χρόνου, να πω ότι καταρχάς θα κλείσω τον κατάλογο των αγορητών. ο τελευταίος και θα περιοριστούμε στο 1,5 λεπτό. Κύριε Δελχάγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω τον εισηγητή, αλλά θα επανέλθω στο θέμα των βιοκαυσίμων. Συμφωνώ μαζί του για την ανάγκη διατήρηση των παροξών επενδύσεων, αλλά αυτό δεν μου φαίνεται συμβατό με τη θέση που είχαμε ή που έχει μάλλον για τα καύσιμα, βιοκαύσιμα πρώτη γενιάς. Να υπενθυμίσω ότι προέρχονται από την κράμβη, από την παραγωγή κράμβης και για την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή θα πρέπει να υπάρχει κάποια ανεξαρτησία σε σχέση με πρωτενε, οι οποίες σήμερα εισάγονται και είναι γενικά τροποποιημένε. Από τη στιγμή που η Ευρώπη δεν έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο για τι πρωτενε στα πλαίσια τη ΚΑΠ στα πλαίσια εξάλλου της ε, κυκλικής οικονομίας έχουμε μια συγκεκριμένη λογική. Δηλαδή από αυτή την γεωργική παραγωγή α πούμε κράμβης εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε πρωτεΐνη και καύσιμα, δύο δηλαδή. Οπότε ακολουθούμε εδώ πλήρως την λογική της κυκλικής οικονομίας και όμως αυτά τα βιοκαύσιμα αποτελούν για τους ε, γεωργούς έναν τρόπο συμπλήρωση των χαμηλών είδη εισοδημάτων τους. Και τέλος, να πω ότι αυτή η έκθεση αφαιρώντας διαδοχικά τα βιοκαύσιμα νομίζω ότι προκαθορίζει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε σχέση με την αθεώρηση της οδηγίας σε σχέση με τις ΑΠΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον ε, κύριο Σόφολη, τον εισηγητή μας. Πρέπει να διακρίνουμε τους διάφορους κλάδους. Στο τέταρτο και πέμπτο πακέτο η Κομισιόν θα πρέπει να έχει ε, κάποιους ε, χαμηλούς συντελεστές ε, συμμόρφωσης. Ε. θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι απαραίτητες ε, προδιαγραφές, ε, παραδείγματος χάρη ε, μετράμε και τις αγελάδες στη χώρα μου, σφάζονται 170.000 αγελάδες κάθε χρόνο λόγω της περιβαλλοντικής πολιτικής. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε συνεχώς και την αφιλία η οποία πλήττεται από την κρίση στον κλάδο του κατηγορουμένου. Θα πρέπει λοιπόν να ε, προτιμούμε τα καλύτερα πλοία, κάτι το οποίο βεβαίως δεν σημαίνει. Υπάρχουν βεβαίως και οι λύσεις όπως το LNG και τα λοιπά και θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αρκετά. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Η ποιότητα του αέρα στην θάλασσα είναι βεβαίως πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε πόλη. Οπότε αυτό το οποίο, στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι οι δρόμοι. Τώρα γιατί κατηγορεί δε και την αεροπορία και τις σχετικούς οργανισμούς ο εισηγητής ότι δεν έχουν κάνει αρκετά δεν είναι κατανοητό ιδιαίτερα αν δούμε το διεθνές πλαίσιο. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπάλτσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκπομπές διο... Ε, αερίων ε, του θερμοκηπίου κατά 25% προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση τέτοιων οχημάτων χρειάζονται τερματικά φόρτισης, χρειάζονται οι σχετικέ υποδομές. Πρέπει όμως να θέσουμε εδώ ένα ερώτημα. Πόσο καθαρή είναι αυτή η ενέργεια που καταναλώνουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, διότι η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα από κάπου προέρχεται. Θα πρέπει να επενέσουμε τη Γερμανία διότι το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας για τα οχήματα αυτά προέρχεται από αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Κατά τα άλλα όμως χρησιμοποιείται ο λιχνίτης. Πολύ σπάνιες είναι οι περιπτώσεις όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρή. Σκεφτείτε ε, τα ποδήλατα που υπάρχουν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών ε, για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων. Αυτή είναι καθαρή ενέργεια, αλλά η ηλεκτρική ενέργεια για τα οχήματα δεν είναι καθαρή. Αν λοιπόν θέλουμε να ε, ενθαρρύνουμε την διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων, θα πρέπει να εξετάσουμε από πού προέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε σαφείς ορισμούς. Θέλουμε καθαρή ενέργεια και η πυρηνική ενέργεια είναι πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε όχι μόνο τις άλλες πράσινες πηγές, διότι και τα πυρηνικά εργοστάσια θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ακούστηκαν διάφορα. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν. Η ε, ε, πολύ ε, σωστά ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα των οξυδίων του αζότου. Θα πρέπει να φροντίσουμε ότι αποφασίζεται να εφαρμόζεται κιόλα. Ε, αν αυτό γινόταν ε, πάντα, τότε θα είχαμε πετύχει πολλά για το περιβάλλον. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Ε, υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία για το Γιβραλτάρα, αλλά αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλά πράγματα. Και επίσης όσον αφορά την ψηφιοποίηση και την οικονομία του επιμερισμού θα πρέπει να φροντίσουμε να στηρίξουμε ε, διάφορες τέτοιες κινήσεις από πλευράς της πολιτικής και να δημιουργήσουμε κίνητρα. Επίσης όσον αφορά την μείωση εκπομπών, αν έχουμε τις ε, κατάλληλες ε, προσφορές ε, τότε θα γίνουν πολλά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα απαραίτητα προγράμματα. Όσον αφορά την υποδομή για τους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά και το υδρογόνο. Η Σουηδία ασχολείται με το θέμα αυτό. Θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά. Ε, βλέπουμε καθυστέρηση όμως ε, στους τομείς αυτούς. Και επίσης, ε, όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, θα ήθελα σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε μείωση των εκπομπών. Αυτό νομίζω θα βοηθούσε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ο τελευταίος ομιλητής μας. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Ζοφόλη, για την γνωμοδότησή του πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ μιλάμε για το μέλλον της κινητικότητας στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε με τρόπο καινοτόμο. Ε, διότι δείτε πώς έχει ρυθμιστεί αυτή τη στιγμή η αστική μεταφορά στην Ευρώπη. Αυτό θα αλλάξει τελείως και μάλιστα εάν το κάνουμε σωστά και προ όφελο όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε αστικές περιοχές. Αυτό ισχύει και για τον καθορισμό των στόχων για την ηλεκτροκινητικότητα. Ε, στόχος είναι να απαλλαγούμε από τις ε, μη αποδοτικές ε, μηχανές εσωτερικής ανάφλεξης στο κέντρο των πόλεων. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αλλάξει απλά εξετάζοντας την αγορά και ελπίζοντας ότι κάπως θα γίνει αυτό από μόνο του. Όλη η υποδομή για τα ορυχτά καύσιμα έχει δημιουργηθεί με υποστήριξη της πολιτικής ήδη από την αρχή και αν θέλουμε να αλλάξει χρειάζονται και εδώ αυστηρές πολιτικές. Και η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με τον καθορισμό των στόχων. Να γνωρίζετε ότι βιομηχανία από μια μεγάλη χώρα που επικεντρώνεται στην ε, παραγωγή μεγάλων αυτοκινήτων, δεν θα αναφέρω τη χώρα, αλλά από γάμα ξεκινάει το όνομά της, Αν ακούσετε κάποιον να λέει ότι ναι, ας έχουμε ε, μείωση των στόχων, να γνωρίζετε ότι μιλάμε για την γερμανική βιομηχανία αυτοκινήτων. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο για πέντε λεπτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ ε, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης μου. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαστε που είμαστε στην συζήτηση αυτή και κοιτάμε και τη συζήτηση που υπάρχει εντό έδωσης. Πρώτα απ' όλα βλέπω πως διαβάστε πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση της Κομισιόν. Ε, περιέχει πολλά πράγματα τα οποία σημείωσαν οι βουλευτές. Βεβαίως αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση και η Κομισιόν έχει πει πως ο γενικός στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του κατά 60% το 2050 σε σχέση με το 1990. Αυτό το 60% πρέπει να γίνει. Ε, αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί κατά 20% οι εκπομπές σε σχέση με το 1990. Οπότε μιλάμε για τεράστια αλλαγή που πρέπει να γίνει. Και στρατηγική, αν θέλετε, ανέφερε τις διάφορες δράσεις που ε, θα έκανε η Κομισιόν τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ε, θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ε, προδιαγραφής διοξιδίου του άνθρακα για αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Με, ε, προετοιμάζουμε προδιαγραφές για μετά το 2020. Θα προσπαθήσουμε να πάμε προς, χαμηλέ, προς οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Η αξιολόγηση αντικτύπου αυτή τη στιγμή εξετάζει το συγκριτικό κόστος και όφελος διαφόρων επιλογών για την αυστηρότητα και τον χρονισμό, οπότε ακριβώ ετοιμάζουμε την πρόταση. Βεβαίω υπάρχει μια απόφαση ήδη για να υπάρξει ο νέος κύκλος δοκιμών που θα τεθεί ενισχύ φέτος και βεβαίω θα προσπαθήσει να μειώσει το κενό μεταξύ των εκπομπών όπως αυτές αναφέρονται και των πραγματικών εκπομπών και βεβαίω θα δούμε και το ζήτημα της επιβολής. Για τα βαρέα οχήματα η Κομισιόν επίσης έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να προτείνει προδιαγραφές στη διάρκεια αυτής της εντολής. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι πιστοποίηση και παρακολούθηση για βαρέα οχήματα και σκοπεύουμε να οριστικοποιήσουμε τις νομοθετικές προτάσεις προσεχώς και κάποιοι βουλευτές ανέφεραν παραδείγματος χάρη τα καθαρά λεωφορεία. Και κοιτάμε ακριβώς τις δημόσιες προμήθειες και το πώς θα βοηθήσουν την κατάσταση. Ε, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή κάνει μια αξιολόγηση αντικτύπου και κοιτάμε ακριβώς ε, την πιθανή αναθεώρηση της ε, οδηγίας. Σκοπεύουμε μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε μια πρόταση για μια πλούστερη και πιο αποτελεσματική ε, λύση. Αναφέρθηκαν επίσης ε, τα οξύδια του αζότου. Όπως ήδη είπε η Επιτροπός Μπιενκόφσκα, η Κομισιόν θα κάνει μια ετήσια ανάλυση των ε, συντελεστών συμμόρφωσης 1 για να φτάσουμε στο συντελεστή συμμόρφωσης 1 για τα οξύδια του αζότου και η εξέταση η φετινή του 2015 θα λάβει χώρα σε μια συνεδρία που θα γίνει 31 Μαρτίου 2017. Για την αεροπορία επίσης ε, πολλά υπόθηκαν. Ε, είμαι σίγουρος ότι ο ΙΚΑΟ στο Μοντρεάλ που ρυθμίζει την παγκόσμια αεροπορία έχει συμφωνήσει σε ένα μηχανισμό αγοράς, ο οποίος θα ξεκινήσει από το 2021, αλλά οι λεπτομέρειες ακόμα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και για τον λόγο αυτόν η Κομισιόν πρότεινε πρόσφατα να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με σταματημένο ρολόι, όπως λέγεται καθώς δεν θα βοηθούσε το να επιβάλλουμε το ETS δεν θα βοηθούσε τις διαπραγματεύσεις και συνεχίζουμε να προτείνουμε σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο το ETS να παραμείνει στο καθεστώς που είχε πέρσι. Και για την ε, ναυτιλία βλέπω το σχέδιο ε, νομοδότησης ε, πως υπήρχε μια πρόταση να μπει η ναυτιλία στο ETS από το 2023. Είναι μια τροπολογία που έχει γίνει στο πλαίσιο και του ETS το θέμα είναι ότι αυτά, τα, αυτές οι δράσεις, δηλαδή το να αποφασίσουμε τώρα το τι θα κάνουμε στο μέλλον, μάλλον ε, δεν βοηθούν στο να έχουμε καλά αποτελέσματα όπως τον, σε οργανισμούς όπως ο ΑΕΜΟ και ο ΕΚΑΟ. Οπότε δεν είμαστε υπέρ του να αποφασίσουμε τώρα. Ας αφήσουμε τους διεθνείς αυτούς τους οργανισμούς να δουν το τι μπορούν να κάνουν και μετά όταν γνωρίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία θα υποβάλουμε τις απαραίτητες προτάσεις. Και τέλος για τα βιοκαύσιμα. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πρόταση οδηγίας ανανεώσιμης ενέργειας. Πέρσι τον Δεκέμβριο προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ παραγωγής βιοκαυσίμων και κάποιων δικλείδων ασφαλείας για να μην δώσουμε κίνητρα, αν θέλετε, για κάποιες ε, ακούσιες συνέπειες ε, της προώθησης ε, των βιοκαυσίμων. Έχουμε λοιπόν ήδη την νομοθεσία που πρέπει να σκεφτούμε. Οπότε αυτή είναι η στρατηγική που σας ανέπτυξα. Υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει το ε, πολύ φιλόδοξο αυτό σχέδιο για να φύγει ο άνθρακας από τις μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής ε, θέλει να πει κάτι σε 30 δευτερόλεπτα. Συνάδελφοι, ευχαριστώ για την συμβολή. Επιβεβαιώθηκε το πόσο ενδιαφέρον και λεπτό και ευαίσθητο είναι το θέμα. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε το στόχο. Κυκλική οικονομία, νέα ανάπτυξη, νέο στυλ ζωής. Η αντίθεση ίσως να αφορά τους χρόνους, τους τρόπους και τα εργαλεία με τα οποία θα φτάσουμε στους κοινούς μας στόχους. Είναι μια πρόκληση που αφορά βεβαίως και τις εθνικές και τοπικές αρχές Πρέπει να υπάρχει και μια συμμαχία μεταξύ βιομηχανίας και περιβάλλοντος για τους διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και κυρίως αυτό να εμπλέκει και τους καταναλωτές, τους πολίτες. Είναι πρόκληση αυτό στην πολιτική, να συγκεράσουμε δηλαδή τους στόχους και τις ιδέες με τους πόρους και την συνένεση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε καλοί και γύρω από αυτούς τους φιλόδοξους στόχους να αναζητήσουμε έτσι μια μακρόπνοη συνένεση για το καλό των δικών μας Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, και Πρόεδρος. Τρεις Μαγιού 11 το πρωί, 29 ψήφος στην Τραν και μετά για τον 5 Σεπτέμβρη επίσης και μετά για την Ολομέλεια θα την έχουμε στη συνέχεια. Επόμενο σημείο. σημείο 12 ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και τον ΕΜΑ σχετικά με τον αντίκτυπο των παράνομων φαρμακευτικών πρακτικών στην υγεία των πολιτών. Η Επιτροπή. Καλησπέρα σας, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με μια μικρή εισαγωγή Τις είπα για τις φαρμακευτικές υπάρχει ένα περιβάλλον που προωθεί τις καινοτόμες ασθενείε, που είναι αποτελεσματικό και υψηλή ποιότητα και ασφαλές. Και το Κοινοβουλίο αλλά και το Συμβουλίο έχουν εκφράσει εμβολίε για τη λειτουργία του φαρμακευτικού συστήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες ασθένειες, σε συγγνώμη θεραπείες. Στο τέλος του χρόνου, η Κομισιόν προετοίμασε μια ανάλυση και αξιολόγησε πρωτοβουλίες. Το SPC, ας πούμε, τα σπιωματικά πιστοποιητικά, για να αξιολογήσουμε ακριβώς τον αντίκτυπο στην πρόσβαση των καινοτόμων θεραπείων. Μετά από την έρευνα λοιπόν, που έκανε η Κομισιόν το 2008-2009, λέει η Κομισιόν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά τις καθυστερήσεις. Η Κομισιόν λοιπόν δημοσίευσε κάποιες εκθέσεις όσον αφορά την εποπτεία των ευρεσιτεχνιών patent και παρόλο που παρουσιάζεται εκεί εν μέρη ε, αυτό το θέμα των προβληματικών ευρεσιτεχνιών, συνεχίζει να παραμένει σχετικά χαμηλό αυτό το πρόβλημα. Πάντως θα πρέπει να δούμε πότε και πώς θα μπορούσαμε να παρανεύουμε όταν ακριβώς έχουμε παράβαση σχετικά με τον ανταγωνισμό. και η Κομισιόν πέρσι τον Ιούνιο τόνισε την ανάγκη ύπαρξη ισορροπίας στα φαρμακευτικά συστήματα στην Ένωση. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις εθνικές αρχές, εθνικές αρμόδιες αρχές και ήδη προετοιμάζεται μία έκθεση όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτής της κατάστασης στους διάφορους φαρμακευτικούς τομείς. Έχουμε το θέμα των δωροδοκιών προς τους ε, γιατρούς, κάτι το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί. Θα πρέπει να εξετάσουμε περιπτώσεις και υποθέσεις ε, και εκτός ε, ένωσης όσον αφορά ας πούμε, τον χρηματισμό αξιωματούχων ΟΣΑ για αυτά τα θέματα. Αν υπάρχει λοιπόν υπόνοια κατάχρηση κονδυλίων της ένωσης από φαρμακευτικές ή φαρμακοβιομηχανίες όλα αυτά θα πρέπει να φέρονται και να μεταβάζονται στην Όλαν. Η Κομισιόν λοιπόν εντόπισε κάποια κρούσματα διαφθοράς και τα ανέφερε στα πλαίσια της, ε, του εξαμήνου για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Επίσης η Κομισιόν δημοσίευσε μια μελέτη το 2013 για αυτό το θέμα, μελέτη η οποία ενημερώνεται συνεχώς διοργάνωσε επίση η Κομισιόν ένα workshop για του εθνικού εμπειρογνώμονε το 2015 για την πρόβλεψη και καταπολέμηση τη διαφθορά σε αυτόν τον τομέα, όπου συζητήθηκε το θέμα τη διαδικασία τη αποφάσεων, του λόμπινγκ κτλ. για αυτού που λαμβάνουν αποφάσει. Τέλο, για τη φαρμακοβιομηχανία, για να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υγεία και στην ευεξία των πολιτών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά οι πραγματικέ ανάγκε που υπάρχουν και το 13 η Κομισιόν διευκόλυνε μία συζήτηση για την ηθική και τη διαφάνεια. Δηλαδή στα πλαίσια αυτό που ονομάζουμε εταιρική υπευθυνότητα όσον αφορά τις φαρμακοβιομηχανίες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε τις αξίες και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και της ηθικής σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους του επαγγελματίε στον τομέα της ε, υγεία και της φαρμακομηχανία. Ελάχιστες προδιαγραφές ε, θα πρέπει να θεσπιστούν και θα πρέπει να προβλεφθούν επίση και ε, διαδικασίε εποπτεία και παρακολούθησης. Είναι ενθαρρυντικό το ότι η βιομηχανία έλαβε υπόψη της αυτές τις αρχές στην χάραξη των δικών της κατευθυντηριών γραμμών όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των αρχών. Αυτά από μένα. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και πρόεδρος. Έχουμε κάποια λεπτά για συζήτηση. Δέκα και κάτι. Ο κ. από την ΕΜΑ. Τρία, τέσσερα, πέντε λεπτά. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην σημερινή συζήτηση. Φυσικά, οι αθέμητες ε, φαρμακευτικές πρακτικές μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, για τους ανθρώπους και φυσικά ε, ο οργανισμός μας ανησυχεί. Αυτές οι αθέμητες πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν τελικά σε μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού, διότι είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη του κοινού και θέλουμε να προστατεύσουμε το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής δουλειάς που κάνουμε. Και θέλουμε επίσης να στηρίξουμε τις καλές προσπάθειες ε, της βιομηχανίας, ε, κάτι που διακυβεύεται ε, με την άπρεπη συμπεριφορά. Πολλά από τα σημεία που προτάθηκαν για τη συζήτηση αυτή ε, είναι θέματα στα οποία δεν συμμετείχαμε άμεσα. Για παράδειγμα, το καθεστώς ε, για την διανοητική ιδιοκτησία και κάποια άλλα θέματα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ωστόσο, θα ήθελα να σχολιάσω κάποια θέματα όπως αυτό της διαφάνειας. Έχουμε βελτιώσει την πρόσβαση στα έγγραφα και ε, τώρα πια δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών με στόχο να αποτρέψουμε και να προλάβουμε ε, αθέμητες ε, πρακτικές. άλλο σημαντικό θέμα όπου έχουμε άμεση συμμετοχή είναι οι επιθεωρήσεις ε, που αφορούν την ακαιρεότητα των ε, δεδομένων και τις ε, καλές φαρμακευτικές και παρασκευαστικές πρακτικές. Η προσέγγιση μας βασίζεται στον κίνδυνο και συνήθως εφαρμόζεται με βάση κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ε, του οποίου λαμβάνουμε γνώση. Όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών, άλλο θέμα που επίσης αναφέρθηκε σήμερα, εμείς ε, δεν έχουμε άμεση επιρροή στη διαμόρφωση των τιμών, αλλά θέλουμε να έχουμε, την, ε, να έχουμε στενή συνεργασία με τους φορείς που διαμορφώνουν την, τις τιμές των φαρμάκων. Θέλουμε η όλη διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική ώστε να έχουμε πιο οικονομικά φάρμακα. Με τη συμμετοχή βέβαια και άλλων ε, πηγών χρηματοδότησης. Αυτά μπορώ να σας πω σε τρία λεπτά. Κάτι στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο είναι η πρόσβαση στα έγγραφα. Έχουμε δημοσιεύσει πάνω από 300.000 σελίδες μέσα στους πρώτους μήνες τα έγγραφα αυτά μπορούν να αποτελέσουν βάση για δημόσιες διαβουλεύσεις σε κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού σε μας. Ένα πράγμα που μας εμποδίζει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα είναι ε, το περιορισμένο προσωπικό μας. Ε, όλα αυτά, δεσμευόμαστε να έχουμε απόλυτη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ε, και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές μας. Η κυρία Σαϊρπίρικ πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αίσθηση στην Ολλανδία και έχουμε τα παράνομα ε, φάρμακα, έχουμε πλαστά φάρμακα και όλες αυτές οι πρακτικές βεβαίως μπορούν να είναι επικίνδυνες. Ε, πάνω από 80.000 ασθενείς ε, το προηγούμενο έτος ε, αναγκαστήκαν να αλλάξουν φάρμακο και αυτό το ανακοίνωσε το Ολλανδικό Ινστιτούτο για την Δημόσια Υγεία με βάση επιστημονικές έρευνες και μετά από τρεις μήνες ένα μεγάλο ποσοστό τους είχε μια μεγάλη επιδείνωση της υγείας του. Αυτά κοστίζουν και στο κράτος και στην κοινωνία πάρα πολλά λεφτά βεβαίως, ε, αλλά και δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα. Και βεβαίως ε, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε, όπως είπε και η συνάδελφος, να προλάβουμε αυτό το ε, ζήτημα και θα ήθελα κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Έχουμε μια συζήτηση που μας υποχρεώνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ακριβείς. Τα φαρμακευτικά εργαστήρια μπορεί να κάνουν καταχρήσεις και αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Αυτό δεν το αφισβητούμε, είναι αλήθεια και είναι κατακριτέο. Είναι στάσεις που θα πρέπει να καταγγελθούν. Μπορεί να έχουμε επίσης και αδικήματα, παράνομες πρακτικές και πρέπει να παρεμβαίνει η δικαιοσύνη και να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι. Αλλά αφού το πούμε αυτό, θα πρέπει να επιμείνουμε στο ότι δεν θα πρέπει, λόγω αυτού του γεγονότος, να βάλουμε στο ίδιο σακί όλο τον κλάδο αυτό και να πλήξουμε ένα ολόκληρο βιομηχανικό τομέα. Είδα, ας πούμε, πώς αντιδράσαμε στην υπόθεση Volkswagen για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τώρα, επειδή υπάρχουν κάποιοι που έτσι, δεν μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι όλη η φαρμακοβιομηχανία τέλο πάντων πλήττει την υγεία των πολιτών. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα να μην τα μπερδεύουμε όλα δηλαδή. Μιλάμε για θέμητες πρακτικές, οπότε θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη διάρκεια της θεραπείας, τη διάρκεια της πατέντας κτλ. Όμως αυτοί οι κανόνες είναι αντικείμενο εποπτείας και θα πρέπει συστηματικά να είμαστε καχύποπτοι γιατί αυτό ε, βλάπτει την καινοτομία. Θα ολοκληρώσω, αλλά νομίζω είναι σημαντικό να το τονίσω αυτό. Τα εργαστήρια λοιπόν είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια λογική κέρδους. Κέρδος όμως που πραγματικά τους επιτρέπει να επενδύσουν μαζικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Αυτά λοιπόν τα κέρδη προσελκύουν τους επενδυτές και τα κεφάλαια που χρειάζονται παρά τους κινδύνους που επιφέρει η πρωτογενής έρευνα. Είναι κέρδη λοιπόν που τους επιτρέπουν επίσης να προσλάβουν και να διατηρήσουν τα καλύτερα τα ταλέντα και εγκεφάλους. Τώρα βεβαίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων θα πρέπει να διασφαλίζει ακριβώ αυτή την εποπτεία σε αυτόν τον τομέα τη φαρμακομηχανία. Όμω να μην τα μπερδεύουμε όλα, γιατί αυτό θα ήταν πολύ κακό για την καινοτομία στον τομέα τη φαρμακομηχανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσουμε σύντομα. Πεντητσίνη. Παρακαλώ, ανάμιση λεπτό μόνο. Πάρα ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Ταραχτήκαμε όλοι φαίνεται όταν είδαμε μια φαρμακοβιομηχανία να πρωταγωνιστεί σε αυτά τα σκάνδαλα, γιατί ο στόχος της πρέπει να είναι η υγεία των πολιτών. Αλλά ας το πάρει το ποτάμι, γιατί αλλιώς θα ζούσαμε εκτός πραγματικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα σκάνδαλα δεν είναι μόνο, δεν θα είναι τα τελευταία και βλέπουμε να υπάρχει ένα διαβολικός ε, συνδυασμό μεταξύ υγείας και κέρδους. Εμεί θεωρούμε ότι αυτά τα δύο πράγματα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα διακριτά, χωριστά. Οπότε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν μπορούμε παρά να κάνουμε μια υποπτία βάσει των αρχών ελέγχου. Οπότε θα ήθελα εγώ να μάθω ακριβώς τι κάνει από αυτού η αίμα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα για το παπυλωμαβύρους έκθεση του 15 της ΕΜΑ που ζήτησε η Δανία και η ΕΜΑ αρνείται οποιαδήποτε σχέση μεταξύ αυτού του εμβολίου και κάποιων συνδρόμων με παρενέργειες. Το Cochrane Center, ένα ανεξάρτητο ερευνικό κέντρο της ε, Νορβηγίας, απευθύνθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ακριβώς για να θίξει το θέμα της ελάχιστη διαφάνειας από την ΕΜΑ σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίε που εκφράζονται όσον αφορά του ε, τους δεσμούς μυστικότητας. Αμφιβολίες σε σχέση ας πούμε με τις ε, πολλαπλές ε, περικοπές όσον αφορά την τελική έκθεση και την επιλογή κάποιων στοιχείων της έρευνας. Οπότε ρωτάω, τι γίνεται με την ομάδα πυρογνωμόνων και στην περίπτωση αυτών των εμβολίων οι χώρες μέλη αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες σε σχέση με τις παρενέργειες. Γιατί φαίνεται ότι η αίμα, στην αίμα μάλλον, πολλοί γιατροί αντιτίθενται με την αναγραφή των παρενεργειών και είναι σαφές ότι αν εμείς ε, δίνουμε μάχη για μεγαλύτερη κάλυψη του εμβολιασμού για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και σαφήνεια όσον αφορά ε, τον εμβολιασμό. Και εδώ νομίζω έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει. Με ευχαριστώ. Η κυρία Καμπεσόν, έχετε το λόγο. Τελευταία μιλήτρια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ξεκινήσω λέγοντας η σχέση μεταξύ καινοτομία και φόβου είναι πολύ επικίνδυνη και στο τέλος χάνει ο ασθενής. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το στοιχείο του κέρδους για να οθήσει μια ισχυρή βιομηχανία, όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό μάλλον να πούμε ότι δεν θα πρέπει υποχρεωτικά αυτό να πλήττει την καινοτομία. Δεν είναι σωστό να το λέμε αυτό. Αναφέρθηκε η έκθεση 2008-2009, όπου η ίδια η Κομισιόν κατέδειξε ακριβώς τις δυσλειτουργίες και το τι έπρεπε να γίνει και είχε ανακοινώσει κάποια μέτρα για το πώς ακριβώς ε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση μέσω συμπληρωματικού πιστοποιητικού κτλ. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω, προβλέπετε να κάνετε μία αναθεώρηση σε σχέση με τα ορφανά φάρμακα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση με αυτά τα φάρμακα όταν έχουμε να κάνουμε με ασθένειες σχετικά σπάνιες και τις τιμές αυτών των φαρμάκων. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε τι γίνεται για τον, με τον, αριθμό, τον υψηλό αριθμό προσφυγών μεταξύ γενώσιμων και πρωτότυπων. Αυτό πώς θα το λύσετε. Θα έχετε μία στρατηγική ας πούμε για την αναβολή της θέσπισης των γενοσύμων μετά για την υπατήτηδα. Τι γίνεται και πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την επανεφάνιση νέων κρουσμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο για απαντήσεις στην αίμα, γιατί πρώτα αναφέρθηκε η αίμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα των ελλείψεων Εμείς έχουμε ένα σχετικά περιορισμένο ρόλο. Δηλαδή στην ουσία θα πρέπει να στηρίξουμε τους ε, εμπλεκόμενους στις χώρες μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων. Τώρα για το άλλο που ρωτήσατε. Ξέρω ότι στον Βορρά της Ευρώπης υπάρχει αυτή η θέση Ξέρω ότι έγινε μια προσφυγή στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Εμείς διαθέσαμε όλο το υλικό μας, τις, τα στοιχεία μας, πληροφορίες μας και μπορώ να σας πω ότι τα συστήματα μας είναι αρκετά εύρωστα. Δεχόμαστε ένα εκατομμύριο ενδείξεων και αναφορών κάθε χρόνο από τις χώρες μέλη και θα ήθελα εδώ να τονίσω το γεγονός ότι ο κάθε ασθενής μεμονωμένα μπορεί να υποβάλει μια αναφορά σε μας. Αυτό νομίζω είναι καλό να το έχουμε κατά νου. Και ο αριθμός άμεσων αναφορών ή προσφυγών των ασθενών, μεμονωμένων ασθενών σε εμά διπλασιάζεται ετησίως. Συζητήθηκε λοιπόν αυτό το υλικό από αυτή την επιχείρηση από το Βορρά και είδαμε ότι υπήρξε κάποια διαφορά κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είναι σαν να καθόμαστε εδώ και εξετάζουμε το τι, μάλλον πάνω στο τι διαφωνούμε. Και αυτό ακριβώς κάναμε με την ε, Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης. Καταλήξαμε λοιπόν στο ότι αυτά τα, αυτό το σύνδρομο δεν έχει γενεσουργό αιτία από το εμβόλιο αυτό. Είναι κάτι το τυχαίο. Δεν είδαμε λοιπόν να υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. 18 εκατομμύρια γυναίκες έχουν εμβολιαστεί και απορρίψαμε ξεκάθαρα το ενδεχόμενο σχέση μεταξύ των δύο φαινομένων. Αυτό που συνεχίζουμε πάντως να κάνουμε είναι να συνεχίζουμε την εποπτεία και την φαρμακοεπαγρύπνηση, ώστε ακριβώς να προωθήσουμε ένα είδο επαγρύπνηση, για το οποίο κάνουμε. Και βεβαίως ε, κάνουμε και αυτές τις εκθέσει αυτές τι μελέτες κάθε χρόνο. Για ε, το HPV, αν δούμε περισσότερε ενδείξει, τότε παρεμβαίνουμε άμεσα. Οπότε απορρίπτουμε τελείως την θέση αυτής της επιχείρησης. συγγνώμη, αυτού του ερευνητικού Ινστιτούτου του Κόχρεϊν. Θεωρώ ότι εντάξει είναι καλό να υπάρχει μια επιστημονική θέση η στάση τέλο πάντων, όμως βλέπω ότι αυτή η θέση δεν έγινε ρεχτή από την επιστημονική κοινότητα. Και μάλιστα είναι διαθέσιμα σε όλους και τα πρακτικά όλων των συνεδριασιών μας. Επ' αυτό ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σας δώσω το λόγο για τρία λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από τις ελλείψεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Το συζητάμε τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Φαρμάκων και των Εθνικών Αρχών Φαρμάκων Γεγονό είναι ότι το φαινόμενο αυξάνεται λόγω των αλλαγών στην λυσίδα διάθεσης που είναι παγκόσμια όπως ξέρετε λόγω των διαφόρων αγορών και του πώς ε, τα φάρμακα φτάνουν στους ασθενείς. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε λύσεις το πώς θα γίνουν, πώς θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Κάποιες χώρες έχουν κάποιες ιδέες που θα ήθελα να μοιραστούν με άλλες και προσπαθούμε να διευκολύνουμε, όπως είπα, μαζί με την ΕΜΕ e και τους επικεφαλείς ε, των ΕΟΦ ε, της, ε, την διαδικασία αυτή, γιατί είναι θέμα και διανομής πρόσβαση στα φάρμακα, αλλά βεβαίω και ένα ζήτημα που σχετίζεται με προβλήματα ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού όταν κάτι παράγεται στην Κίνα ή στην Ινδία μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση στα φάρμακα. των ασθενών. Οπότε ε, δεν θέλω να πω ότι θα βρούμε ε, λύση γιατί δεν υπάρχει κάποια εύκολη λύση. Έχουμε και τις νέες πληροφοριακές λύσεις που έρχονται. Απλά θα προσπαθήσουμε ακριβώ να υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ε, ειδοποίησης ο οποίος θα λειτουργεί γρηγορότερα. Έχουμε και την Προεδρία της Εστονίας η οποία θα οργανώσει μια σχετική συνάντηση για την έλλειψη των φαρμάκων και μια νέα ψηφιακή προσέγγιση. Για να απαντήσω σε ερωτήσεις κυρία Καβάζα γιατί ότι συνέχεια θα δοθεί στις ε, περιπτώσεις ε, που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού. Όπως είπα, η Κομισιόν συντάσσει αυτές τις εκθέσεις για την εφαρμογή των πρακτικών αυτών. Ταυτόχρονα έχουμε κάποια ζητήματα δικαίου του ανταγωνισμού Έχουμε τρεις τέτοιες περιπτώσεις, η τέταρτη έκρεμη η απόφαση πέρσι τον Σεπτεμβρίου του δικαστηρίου ε, βεβαίωσε την απόφαση της ε, Κομισιόν, κάτι το οποίο σημαίνει ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ακριβώς ε, αυτά τα οποία κάλυπτε η μελέτη για την υπόλοιπη τη νομοθεσία. Προσπαθούμε να τι γίνεται. Να ολοκληρώσουμε την έκθεση με κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζουμε να σας παρουσιάσουμε κάποιες εκθέσεις για τα παιδιατρικά φάρμακα φέτος και να δούμε τα προβλήματα στον τομέα αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα και συνεχίζουμε αμέσως με το σημείο 13 το οποίο αφορά δημόσια ακρόαση σχετικά με τα πρόσθετα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Και χαίρομαι που καλωσορίζουμε πέντε εξωτερικούς ομιλητές. Οπότε στόχος είναι να γίνει ένας απολογισμός και να τονίσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την δημοσιογεία των πολιτών μας. Για όλους μας ε, είναι σαφές. Αλλά για πολλούς πολίτες της Ένωσης το ζήτημα αυτό παραμένει ανοιχτό και κάτι πρέπει να κάνουμε για να το επιλύσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον κύριο Πίτερ Ντεπό Πριντάν Ελκ και για τους υπόλοιπους ομιλητές παρακαλώ να περιοριστείτε σε 10 λεπτά στις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να είμαστε εδώ. Ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας για τα επιτεύγματα και το τι έχει επιτύχει μέχρι στιγμής η περιβαλλοντική πολιτική. Τι βεβαίως εμείς είμαστε, είναι ασυνήθιστο αυτό για εμάς γιατί είμαστε περιβαλλοντική μοικείο, αλλά θεωρούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα απολογισμός Λοιπόν υπάρχουν τρεις ε, κύριες ε, προτεραιότητες. Συγγνώμη. Για να ε, βρω λίγο εδώ το κουμπάκι. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν έχουμε στο έβδομο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο. Το ένα είναι η φύση και η βιοποικιλότητα. Κοιτάξτε, με βάση τις πολιτικές ε, της Ένωσης ε, έχουμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Ένα ολόκληρο φάσμα ειδών που ε, επανεμφανίζονται ενώ κόντευαν να εξαφανιστούν. Τα πάλι το παράκανα. Παραδείγματο χάρη τα αποδημητικά πουλιά. Πλέον δεν σφάζονται αδιακρίτως στο νότο της Ευρώπης. Εδώ έπαιξε ρόλο το Life Fund για να μην εξαφανιστούν ήδη όπως ο Λίγκας της Σιβηρικής και η οδηγία περί και βιοτόπων που έχουν ήδη αρχίσει να αναστρέφουν την κατάσταση των σημαντικότερων ειδών και βιοτόπων. Και από ό,τι φαίνεται δημιουργούν ε, και κέρδη, ωφέλη 9 ε, εκατομμυρίων ευρώ κατ' από τον τουρισμό. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν που δεν θα είχαν συμβεί χωρίς τις πολιτικές της Ένωσης. Το ίδιο βλέπουμε και στον τομέα της καθαρής ε, κυκλικής οικονομίας, συνδυασμός δηλαδή δεσμευτικών στόχων και μέτρων μέτρων στήριξης για ανανεώσιμες αποτελεσματικότητα ε, που μετατρέπουν ε, τον τομέα της ενέργειας σε πάροχο υπηρεσίας. Δηλαδή αντί να πουλάνε κιλοβατόρες, ε, πουλάνε μια υπηρεσία. Ευθυρότερε προδιαγραφέ διοξιδίου του άνθρακα που έχουν εγκριθεί για αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά έχουν βελτιώσει την κατανάλωση καυσίμων, την ποιότητα του αέρα και έχουν αλλάξει και τη βιομηχανική στρατηγική των μεγάλων κατασκευαστών ε, που ε, βεβαίως απομακρύνονται από το δίζελ. Και βεβαίως ε, φεύγουμε από μια γραμμική και πηγαίνουμε προς μια κυκλική οικονομία. Όλα αυτά λόγω των πολιτικών, των προσπαθειών που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα και ο οικολογικός σχεδιασμός και η ενεργειακή σήμανση ε, που είχαν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 6.900 ε, πέτατζάουλ ενέργειας. 336 ε, εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού και εξοικονόμηση 112 δισεκατομμυρίων ευρώ από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης, στον τομέα της υγιεινής και της ε, ασφάλειας ε, και εκεί πέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν θα συνέβαιναν χωρίς αυτές τις προδιαγραφές. Παραδείγματος χάρη ε, τα πλαφόν για νέονεκ ή το ότι την Παρασκευή θα εγκριθούν νέες προδιαγραφές για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης παρά το ότι απειλεί η Γερμανία πάλι θα μειώσουν ε, τον αριθμό πρόωρων θανάτων από 20.900 σε 2.600 στον τομέα των χημικών ουσιών. Ο κανονισμός REACH ε, σημαίνει ότι ε, προχωράμε σε μια υποκατάσταση επικίνδυνων χημικών ουσιών, ποτάμια και παραλίες καθαρίζουν, η ρήπανση με βαρέα μέταλλα, με φόσφορο, επικίνδυνες χημικές ουσίες ε, έχει αρχίσει να μειώνεται κατά πολύ και για να έρθουμε λοιπόν στο τι είναι η προστέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, όταν 28 κράτη-μέλη, 28 ακόμα είναι, ε, συνεργάζονται με ένα κοινό στόχο για το πώς θα κάνουν τα πράγματα και έχουν ε, μετρήσιμα κριτήρια, μιλάμε για μια τεράστια διαφορά και κάνουμε πράγματα από κοινού που δεν θα μπορούσε να κάνει ο καθένας μόνος του. Να το. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση de facto γράφει κανόνες του κόσμου. Και... Νομίζω πως ε, έχουμε ένα μοναδικό ρόλο και έτσι υπάρχει καινοτομία, επενδύσεις και βεβαίω η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει το πλέον έκτημα του ότι ε, κινείται πρώτη βεβαίω, Ταυτόχρονα ε, έχουμε και ίσους όρου ανταγωνισμού εντό τη Ένωση και κατ' ουσίαν αυτό μας επιτρέπει να δούμε τις διασυνοριακές επιπτώσεις της ρήπανσης και άλλων πιέσεων και των καθαρών περιβάλλων ε, είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες και το βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι πρόκειται για έναν τομέα όπου γενικά οι πολίτες θεωρούν ότι πρέπει να κάνει και περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι λιγότερα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιους κινδύνους όμως και ευκαιρίες, γιατί υπάρχει μια επιτυχία μεν, αλλά βεβαίως ως περιβαλλοντική μοικείο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Παραδείγματο χάρη απειλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ρόλο της ε, ε, λόγω της ε, κακής εφαρμογής. Επίσης υπάρχουν ζητήματα όπως η καλύτερη νομοθεσία και τα ζητήματα του εμπορίου όπου βλέπουν την ρύθμιση αυτών των θεμάτων ως εμπόδιο, ως βάρος και δεν βλέπουν την περιβαλλοντική πολιτική ως ένα μέσο το οποίο μας βοηθάει για να λύσουμε κάποια από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε. Ταυτόχρονα έχουμε μια παγκόσμια ατζέντα με τους αναπτυξιακούς στόχους ε, τους 17 στόχους που έχουμε που είναι νομίζω μια, ένας πολύ καλός στόχος και θα ήθελα να ολοκληρώσω με τις προοπτικές για το 2030. Πρώτα απ' όλα. Μπορούμε να πούμε ότι η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πετυχημένη. Η δήλωση της Ρώμης πριν από λίγες εβδομάδες ήταν ένα μήνυμα πολλά υποσχόμενο. Δηλαδή αναγνώρισαν οι ηγέτες ότι το καθαρό περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το μίσο που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται και πρέπει να συνεχίσει αυτό. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε όλα όσα έχουμε κάνει. Ε, δεν αρκούν, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Στην κλιματική αλλαγή πρέπει η μετάβαση να γίνει πολύ πιο γρήγορα σε όλους τους κλάδους, ειδικά στον τομέα της γεωργίας, αεροπορίας, ναυτιλίας, ε, να περάσουμε στις προδιαγραφές και για τα φορτηγά, όχι μόνο τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά. Βιοπικιλότητα, ρήπανση των υδάτων, πολλά από αυτά προέρχονται από τη γεωργία. Πρέπει να υπάρξει και μια αλλαγή στη γεωργία. Και να αρχίσουμε να κλείνουμε το κενό εφαρμογής που υπάρχει. Να αρχίσουμε να αυστηροποιούμε τις προδιαγραφές. Π.χ. θα ψηφίσετε π.χ. όρια για το κάδμιο στα λοιπάσματα. Αυτό πρέπει να το βάλετε στα 20 μιλιγκράμμ. Τέλος. Για να κοιτάξουμε και λίγο στο μέλλον το θέμα της πολιτικής συνέχειας. Έχει μεγάλη σημασία και βλέπουμε ακριβώς τα προβλήματα της ασυνέχειας όταν α, ε, ε, εσείς ρωτήσατε τον Επίτροπο Βέλα, είπατε ότι ήταν καλός για δουλειά, κλείνωσε μια νέα εντολή, την οποία τελικά δεν έλαβε. Πηγαίνουμε λοιπόν προς νέες ευρωεκλογέ νέα κομισιόν, πρέπει να ξεκινήσουμε το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον, να υπάρχει μια συνέχεια πάνω σε αυτό το θέμα, οπότε ε, εδώ τελειώνω και σας ευχαριστώ και πάλι. Thank you, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, καθώς και για την νότα αισιοδοξία ε, στο τέλος της παρέμβασής σας, ε, διότι ο επόμενος ο μιλητής μας, ο Τόντ Στέρν, ήταν αρμόδιος ε, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ήταν και ο κύριος διαπραγματευτής της κυβέρνησης Ομπάμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Μ' ακούτε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, για την πρόσκλησή σας να εμφανιστώ εδώ σήμερα. Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα ε, ε, ε, επιμέρους συναντήσεις με τους ευρωβουλευτές. Σήμερα όμως είναι η πρώτη μου δημόσια εμφάνιση. Μου ζητήθηκε να αναφερθώ στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και να σας πω ήδη από την αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο πιο σημαντικός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πάνω από 7 χρόνια της θητείας μου ως ειδικό απεσταλμένου του Προέδρου Ομπάμα. Δεν ε, συμφωνούσαμε πάντα σε όλα τα θέματα, συμφωνούσαμε όμως όσον αφορά τα θεμελιώδη θέματα. Ε, το πόσο απαραίτητο ήταν να ε, καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος με τρόπο προορατικό. Στις περιπτώσεις όπου διαφωνούσαμε, η κοινή μας δέσμευση να πετύχουμε το στόχο μας και η κοινή μας οπτική μας επέτρεπε να βρούμε κοινό τόπο. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι το εξή, ότι δεν θα υπήρχε ε, η ιστορική συμφωνία του Παρισιού χωρίς ε, την μοναδική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ζωτικό ρόλο ε, συχνά κάναμε δύο βήματα μπροστά και ένα και τρία τέταρτα βήματα πίσω, αλλά πάντα προχωρούσαμε μπροστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα σταθερή και αξιόπιστη. Δεν είναι κρυφό ότι η πολιτική κατάσταση όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος ε, ήταν ε, πολύ πιο ασταθής στις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την, τις απόψεις του κοινού στο θέμα αυτό στη, στις Ηνωμένε Πολιτείες και έχω ελπίδες και για το μέλλον. Ωστόσο, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σταθερότητά της ήταν πολύ χρήσιμη τα τελευταία χρόνια. Πάντα γνωρίζαμε και ο κόσμος όλος γνώριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούσε, ήταν αξιόπιστη και ότι παρέμενε δεσμευμένη να πετύχει τους στόχους όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν μια ισχυρή φωνή για φιλόδοξες συνομιλίες για το κλίμα. Πάντα επιχειρηματολογούσε, ε, ήθελε φιλόδοξους στόχους ε, καθώς ε, και εξέταση κάθε πέντε χρόνια ε, σχετικά με το αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Μάλιστα, κατά τις διαπραγματεύσεις του 2011, στις διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν στον Τέρβαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε να δημιουργηθεί συνασπισμός χωρών που ζητούσαν δράση φιλόδοξη και μια νέα συμφωνία που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε και μετά το 2020 θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στην Κοπενχάγη και στην Κανκούν το 2009 και 2010 αντίστοιχα είχαμε διαπραγματεύσεις. Ε, κάλυψαν όμως το, διάστημα μόνο μέχρι το 2020 και ενώ ήταν ε, μια σημαντική αρχή δεν ε, προχωρούσαν αρκετά. Στο Ντέρμπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σειρά άλλων χωρών συμφώνησαν να έχουν πιο φιλόδοξους στόχους. Και έτσι στο Τέρπαν ε, είχαμε μια νέα εντολή για διαπραγμάτευση της νέας συμφωνίας, ε, τη λεγόμενη πλατφόρμα του Τέρπαν. Τέσσερα χρόνια αργότερα και οι Ηνωμένε Πολιτείε συμμετείχαν στο συνασπισμό αυτόν... και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού. Μπορεί να είμαι ο πρώτος που χρησιμοποίησα τον όρο συνασπισμός υψηλής φιλοδοξίας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση το πέτυχε αυτό και δεν ε, θα υπήρχε συνασπισμός ε, για διεύρυνση των συζητήσεων το 2015 αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε βοηθήσει στη δημιουργία του συνασπισμού αυτού το 2011. Η φύση της Συμφωνίας του Παρισιού από τη βάση προς τα πάνω και ξεκινώντας από το εθνικό επίπεδο, αυτή η προσέγγιση ήταν πολύ χαρακτηριστική. Αλλά μια καλή αρχιτεκτονική, μια καλή δομή δεν μπορεί να περιορίζεται στη βάση. Και η σημασία της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καταστάθηκε ικανή λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία συμμαχία πολλών χωρών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τι χώρε του Βορρά, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και άλλου. Όλε οι χώρε αυτέ έχουν συμβάλει σημαντικά. Αλλά ε, μην ε, απατώμεθα, η ισχύ και η επιρροή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τέτοια που δεν μπορεί να την φτάσει κανένα μεμονωμένο κράτος. Ήταν πολύ δύσκολο να συντονιστεί η πολιτική τόσων διαφορετικών χωρών. Ε, συχνά είχα και εφιάλτες σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά το αποτέλεσμα το να, το να μπορώ να συνομιλώ με μία ενιαία ομάδα ε, ήταν πολύτιμη. Να κλείσω λέγοντα το εξής. Ε, το θέμα της Συμφωνία του Παρισιού δεν έχει λήξει. Χρειάζονται πιο αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορους τομείς, ε, μεταξύ άλλων ε, για την διαφάνεια, που προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2018. Επίσης, προβλέπεται ένας διάλογος διευκόλυνσης που θα ξεκινήσει με μια εξέταση της κατάστασης για να εξεταστεί το κατά πόσο πληρούν ε, οι συμβαλόμενες χώρες τους στόχους και επίσης θα έχουμε μια σειρά ε, κύκλων ε, πέντε ετών. Υπάρχουν κάποιοι που δεν ήθελαν την συγκεκριμένη ισορροπία που πετύχαμε ήδη από την αρχή και πολύ ευχαρίστω θα οπισθοχωρήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας να θυμάστε ότι η Συμφωνία του Παρισιού κατέστη δυνατή μόνο και μόνο επειδή πολλές διαφορετικές χώρες και ομάδες χωρών με πολύ διαφορετικές οπτικές ε, κατέληξαν σε δίκαιους συμβιβασμούς. Δεν επιτρέπεται πια να οπισθοχωρήσουμε από αυτά που πετύχαμε στο Παρίσι. Θα κλείσω εδώ. Με εκπλήσει το γεγονό ότι δεν χρησιμοποίησα όλο το χρόνο ομιλία μου, πάντω ευχαρίστω θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σημαντικό αυτό που μα είπατε. Ήσασταν από τους διαπραγματευτέ. Θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Δημοσιαγία. Νίνα Ρέτσο είναι ο κύριος συγγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα για το σημαντικό αυτό θέμα. Θα συνεχίσω με το θετικό πνεύμα της ακρόασης και να θα πω ότι η σύμβαση για την υγεία είναι, η συνθήκη για την υγεία είναι νέα, νεαρής ηλικίας, 25 αλλά ξεκίνησε από το 80 όταν η Ευρώπη συμμετείχε στην καταπολέμηση του AIDS και της κατάξυσης ναρκωτικών. Έχει λοιπόν η Ευρώπη ένα σημαντικό βαθμό επιδόσεων όσον αφορά τα θέματα αυτά. Αυτός ο, αυτές οι επιδόσεις βεβαίως μας καθοδηγούν και νομίζω ότι η, Ευρω... υγεία είναι από τα μεγαλύτερα success story της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προσβλέπουμε και σε περαιτέρω μελλοντικέ επιτυχίες. Να πω καταρχάς ότι έχουμε τις εθνικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο ως σύστημα υγείας εθνική αρμοδιότητα και μεταξύ των διαφόρων φορέων νομίζω ότι κανείς δεν ζητάει μια ενιαία αγορά υγείας, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική υγείας, οπότε αυτό θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Όμω του λεχθέντος, εκεί που η Ένωση έχει αρμοδιότητα για να δράσει, είναι η συμβολή στην λειτουργία, συνέχιση και βιωσιμότητα όλων των εθνικών μας συστημάτων για στην Ένωση. Μακροοικονομική, βεβαίως ευρύτερα. Και θα εξηγήσω το γιατί. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση πέτυχε πολλά για τις υπηρεσίες υγείας μας και για την παροχή σημαντικών πόρων. Είχαμε ασφαλή φάρμακα, ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών, ε, εξοπλισμό. Είναι βέβαιο, ας πούμε, ότι αν θα χρειαστείτε μετάγγιση αίματος εκτός, εκτός χώρας σας θα το έχετε και ότι έχετε πρόσβαση τέλο πάντων στα φάρμακα που χρειάζεστε. Αυτό χάρη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χάρη στα δικαιώματα και στην προστασία που παρέχουν τα εθνικά συστήματα. Έχουμε και προϊόντα βέβαια, τα οποία παραμένουν βλαβερά για την υγεία μας, αλκοόλ, καπνός κτλ. Έχουμε και ένα είδος ελεύθερης κυκλοφορίας άλλου είδους, δηλαδή μικρόβια, μικρόβια που είναι αθεκτικά στα φάρμακα κλπ. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς βεβαίως ε, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και δηλαδή προστασία κατά αυτών των απειλών. Η Ευρώπη έχει μακρά ιστορία αντιμετώπισης αυτών των απειλών και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, καρκινογόνα, οδικά ατυχήματα και πολλά πολλά άλλα. Πάρα πολλά από αυτά αντιμετωπίστηκαν και σε τομείς εκτός υγείας, στις μεταφορές, στη γεωργία, στο περιβάλλον. Η νομοθεσία και οι συνθήκες συνήθως ακολουθούν την επιδημιολογία αργότερα. Και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα όπου εδώ το κοινοβούλιο ήταν σημαντικό σε κάποιες πολιτικές υγείας. Καταρχάς, ο έλεγχο του καπνίσματος. Το υπάρχον πλαίσιο επέτρεψε στις χώρες να προχωρήσουν πολύ πέραν ε, αυτό που θα είχε επιτρέψει το λόμπι του καπνού. Πριν κάποια χρόνια ήμασταν στο 50% άρων καπνιστών στην Ευρώπη. Έχουμε πέσει τώρα κάτω από το 30% και αυτό μέσω διαφορών πολιτικών που άλλαξαν και μείωσαν το ποσοστό καπνιστών και του θανάτους αντίστοιχα. Σώσαμε λοιπόν ζωέ και ελαφρύναμε και το βάρος στα συστήματα υγεία μας. Συνεχίζουν να μειώνονται λοιπόν οι αριθμοί των καπνιστών ετησίω, αλλά συνεχίζουμε να σκοτώνουμε 700.000 ε, άτομα ετησίω. Κάθε δευτερόλεπτο περνάει θα πεθάνει πρόωρα κάποιο καπνιστή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα διεύρυνε και την επιρροή της παγκοσμίω επειδή πρωτοστάτησε στον έλεγχο του καπνίσματος. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένα, μια συνθήκη που υπογράφηκε από 180 χώρε παγκοσμίω και έσωσε πολλέ ζωέ. Μετά, πολιτικέ για την ασφάλεια την οδική. Είχαμε ένα στόχο μείωσης μέχρι το 2010 κατά το ίμιση των οδικών ατυχημάτων και των θυμάτων. Το πετύχαμε σχεδόν με 43% μέσω θέσπισης προτύπων, μέσω δαπάνης στην υποδομή και βεβαίως χάρη στην εφαρμογή και θέση ισχύ εθνικών μαθησιών που αφορούν τη ζώνη ασφαλείας, ε, το, τον αλκοολισμό κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι πώς όλα αυτά μπορούν να πετύχουν όταν παντρεύουμε ακριβώς λοιπόν εθνικές και ευρωπαϊκές ε, πολιτικές, κάτι που ήταν πολύ αποτελεσματικό. Πολιτικές για την ποιότητα του αέρα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Κατά ένα τρίτο μειώθηκε, μειώθηκε ο αντίκτυπο των οδικών μεταφορών, επίση τη αεροπλοεία κτλ. Είχαμε πολύ, πολύ ψηλά ποσοστά. Βεβαίω έχουμε και άλλα στοιχεία και εξελίξει στο Dieselgate, το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε και να αποπτεύσουμε και σα ευχαριστώ βεβαίω που μα στηρίξατε σε αυτό. Και πάλι πρέπει να σα πω ότι μένουν πολλά να γίνουν. Τα σωματίδια τα οποία προκαλούν 400.000 πόρου θανάτου ετησίω και έχουμε 900 δις ως αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία, οπότε κάθε πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό. Γι' αυτό ακριβώ του λόγου είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που δεν περιλαμβάνει την προστασία της υγείας των πολιτών και των καταναλωτών. Η υγεία και η υγιής οικονομία σχετίζονται άμεσα. Το προσδόκιμο ζωής και η διατήρηση και αύξησή του νομίζω βοηθά την οικονομία. Κατά 4% του ΑΕΠ έχουν υπολογίσει. Έχουμε επίσης και το 5% το οποίο προβλέπεται μέσα TTIP, οπότε θα πρέπει να καθορίσετε γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να θεωρήσει προτεραιότητε τη. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλε αποκλήσει μεταξύ χωρών ε, που θα πρέπει παρόλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει ας πούμε στο προσδόκιμο ζωής διαφορά δεκαετών μεταξύ Ιταλίας και Λιθουανία και τα παραπάνω χρόνια δεν είναι απαραίτητα πιο υγιή. Μπορεί κανείς να ζει περισσότερο δηλαδή, αλλά δεν ζει πιο υγιή. Μπορεί να έχει α πούμε χρόνιε παθήσει. Η στρατηγική της Λισαβόνα ζήτησε την επίτευξη δύο παραπάνω υγιών ετών ζωής, αλλά δεν θα το πετύχουμε, παρόλο που θα έχουμε μια στρατηγική για τι χρόνιε παθήσει, για διαβίτη καρκίνο κτλ αλλά ακόμα δεν έχουμε δει ούτε καν προσχέδιο αυτής της ε, στρατηγικής και βέβαια δεν θα πετύχουμε αυτό τον στόχο, κάτι το οποίο βέβαια θα κοστίσει πολλά δις ε, στα εθνικά συστήματα. Θα ήθελα τώρα να τονίσω το θέμα της ισότητας για την υγεία. Υπάρχει, υπάρχουν 20 χρόνια διαφορά στη διάρκεια ζωή μεταξύ των πιο προχωρημένων και των πιο και των χειρότερων περιοχών τη Ευρώπη από αυτή την άποψη. Ας πούμε για τους Ρωμά υπάρχει πολύ κακή εικόνα. Οι γυναίκε με πεθαίνουν στα 43, οι άστεγοι στα 47, λόγω ακριβώς των πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, θέματα υγείας, θέματα πρόσβασης στις δομές υγείας κλπ. Έρευνα για την υγεία, δεν το ανέφερα αλλά θα ανακύψει στη συνέχεια η προσθέμενη αξία τη ε, διεθνού έρευνα για την υγεία παγκοσμίω είναι ανεκτήμητη. Όχι μόνο σε σχέση με τα μηχανήματα και τι τεχνικέ και του εθνικού προπολογισμού τα συστήματα υγεία, αλλά για την γενικότερη υγεία σε σχέση με την απασχόληση και την εκπαίδευση. Αυτό που δεν έχουμε κάνει αρκετά καλά μέχρι τώρα είναι το να μεταφέρουμε ακριβώς τη γνώση από τα πειραματικά προγράμματα στην Ένωση στις ε, διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονται και λυπάμαι που και το Brexit δυστυχώς παρέχει δυνατότητα για ένα φυσικό πείραμα να δούμε το πώς ακριβώς, ε, τι ακριβώς αξίζει η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για μια χώρα. Και η φυγή εγκεφάλων έχει ήδη ξεκινήσει. Όμως, όλοι θα χάσουμε αν ακριβώς θα χάσουμε την, τις δυνατότητες που παρέχει το νούμερο Βασιλείο σαν αφορά τη συνεργασία στα θέματα αυτά η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να προσέξει ώστε φεύγοντα από την Ένωση να μην πλήξει του ασθενεί και του πολίτε περαιτέρω. Ξέρουμε πολύ καλά το πώ δουλεύουν αυτέ οι πολιτικέ και σε ποιου τομεί οι χώρε θα ε, πάνε καλά συγκριτικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τα πάει καθόλου καλά όσον αφορά του πρόωρου θανάτου και το screening για τον καρκίνο και την πρωτογενή ε, εκεί θεραπεία θα πρέπει να, να υπάρξουν βελτιώσεις εδώ. Και κάποια τελευταία σχόλια. Ένα το ότι, όπως είπε το Ευρωβαρόμετρο για το Κοινοβούλιο πέρσι, γύρω στις 30.000, ε, θέλουμε ε, εμείς να κάνει περισσότερα η Ένωση στον τομέα της υγείας, να αναγνωρίσει τις ανησυχίες που υπάρχουν και να ενισχύσει τις δομές υγείας. Αυτό θα ήταν πολύ καλός τρόπος επαφής με τους πολίτες, δηλαδή ώστε να δει κάθε πολίτης τι κάνει για αυτόν και την οικογένειά του η Ένωση. Τέλος, να πω ότι τα πράγματα της Ένωσης έχουν σώσει πάρα πολλές ζωές. Δεν ξέρουμε πόσα, πόσα επιδημίες γλιτώσαμε, πόσα, πόσα ατυχήματα στον δρόμο, πόσους καπιστές πείσαμε να σταματήσουν το τσιγάρο. Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές σώσαμε. Και θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε τις επιτυχίες μας αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες μας στις χρόνιες παθήσεις, στην ψυχική υγεία, στο AIDS, στη θυματίωση, ε, στην παξαρκία. Χάρη ίσως στις ε, επιτυχίες μας για το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή έγινε το πρώτο αιτίο θανάτου. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με την ε, αντίσταση αντιβιωτικά. Και αυτή είναι η καλύτερη στιγμή ακριβώ για να συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε την υγεία μας. Νομίζω ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 10 εκατομμύρια θανάτους από ασθένειε που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντιβιωτικά. Και πολλές φορές είναι σε χώρες που θεωρούν δεδομένα τα υψηλής ποιότητα συστήματα υγείας. Το καλό νέο είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια που ανέφερα προηγουμένως μπορούν να αποφευθούν διαβήτης κτλ. Νομίζω ότι η ανάπτυξη στόχων μας παρέχει ακριβώς τα εργαλεία και τους τρόπους μέχρι να για να φτάσουμε εκεί μέχρι το 2030. Τώρα θα πρέπει διεθνώ το θεματολόγιο να τα περιλάβει αυτά. Το G20 το, G20 συζήτησε και ο ρόλος της Ευρώπης είναι απαραίτητος. Θα πρέπει όλα αυτά να τοποθετηθούν ψηλά στο θεματολόγιο και σας ευχαριστώ όλους που μας ε, βοηθήσατε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Συνεχίζετε να κάνετε έτσι να φασαρεί για αυτά τα θέματα, να μας βοηθήσετε περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ο κύριος Κιτοράση, ο διευθυντής. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, μας τιμά που είναι η πρώτη υπηρεσία που λαμβάνει τον λόγο τώρα. βεβαίω θα σα παρουσιάσω την σκοπιά του EMA που νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα το φέλους της νέας αγοράς. γιατί πραγματικά παρέχουμε ένα ενιαίο περιβάλλον για υψηλή ποιότητα και ασφαλή φάρμακα προ όφελο των ασθενών, τη πανεπιστημιακή έρευνα και των επιχειρήσεων. Ενία λοιπόν αξιολόγηση, αγορά και ασθενεί. Με το email λοιπόν μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα δηλαδή αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη προστεθέμενη αξία όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Εμείς έχουμε ένα ενιαίο, μια ενιαία δεσμή κανόνων και προτύπων και η σύσταση μας προς την Κομισιόν πριν την τελική έγκριση φαρμάκων, αποδέχεται, ή μάλλον είναι αποδεχτή σε όλη την Ένωση. Έχουμε πιστοποιημένου, εμπειρογνώμονες, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ήδη κάποιου εμπειρογνώμονε που έχουν ελεγχθεί για αντικρώμενα συμφέροντα, για και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσφύγουμε σε αυτούς δηλαδή για να στηρίξουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Αυτό είναι ένα μοναδικό νομίζω περιβάλλον. Η Ευρώπη έχει ωφεληθεί από, από αυτό το τεράστιο δυναμικό τροφοδότησης πραγματογνωμοσύνης και νομίζω ότι εμείς θα μπορούσαμε να ήμασταν πολύ περήφανοι γι' αυτό. Το δεύτερο όφελος είναι ότι, ότι αυτό το εύρωστο σύστημα, όπως είπαμε σήμερα, μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε και να επαπτεύσουμε την ασφάλεια των ε, φαρμάκων μετά την αδειοδότηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή πολλές φορές έχουμε κάνει διαφορετικά συστήματα και διαφορετικά περιβάλλοντα, πέρα δηλαδή των κλινικών δοκιμών. Αυτό έχει άμεση σημασία για τους ασθενείς. Επίσης, στηρίζουμε την καινοτομία, συνεχίζοντας τις προσπαθειές μας, ώστε αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο ισχυρές. Και για να βοηθήσουμε τους ερευνητές και τους επιστήμονες, ώστε να παράξουν περισσότερα και πιο αποτελεσματικά επιστημονικά στοιχεία. Η Ευρώπη λοιπόν είναι στην ε, πρωτοπορία όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές και νομίζω ότι η ανάλυση ωφέλους κινδύνου είναι ακριβώς κάτι το οποίο λαμβάνει ισχυρά υπόψη του το παράγοντα τιμή. Για να καταλήξω, θα ήθελα να πω ότι για να τα πετύχουμε όλα αυτά βασιζόμαστε στη διαφάνεια, που αποτελεί τον ακρογωνίο λίθο μας και το πιο ισχυρό εργαλείο για να οικοδομήσει κανείς αξιοπιστία, να πετύχει εμπιστοσύνη και για να συνεχίσει να λειτουργεί και να προωθεί την ε, επιστημονική καινοτομία. Δεύτερος πυλώνας είναι βέβαια η φαρμακοαπαγρύπνηση και ασφάλεια των φαρμάκων. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και για να συνοψίσω σύντομα να σας πω ότι έχουμε τρεις πηγές πληροφοριών επαγγελματίες υγείας, επιχειρήσεις ασθενείς συν κάποιες μελέτες τις οποίες κάνουμε όταν έχουμε αφιβολίες. Έχουμε λοιπόν και απολαμβάνουμε ενός από τα πιο ισχυρά συστήματα στον κόσμο. Προσπαθούμε λοιπόν να κατευθύνουμε τους παραγωγούς φαρμάκων προς τις ιατρικές ανάγκες και όχι μόνο προς τις ε, ευκαιρίες κέρδους και προσπαθούμε η καινοτομία να φτάσει στους ασθενείς έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να ε, ασκούμε τις υποχρεώσεις μας ε, χωρίς τους οργανισμούς. δίνω τώρα τον λόγο στον Ανδρέα Αμμόν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο, στην κυρία Αμών, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τον Μάιο του 2005 ξεκίνησε τις λειτουργίες του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στην, Σουηδία, στην πρωτεύουσα της Σουηδίας. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένας οργανισμός που ασχολιόταν με την παρακολούθηση των νόσων στην Ευρώπη. Στόχος ήταν να εξετάσει και να εντοπίσει κινδύνους ε, από νόσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύοντας έτσι την υγεία όλων όσων μένουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είχαμε το SARS ε, τον Φεβρουάριο του 2003 και είδαμε πολύ γρήγορη εξάπλωση του ιού αυτού στον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Και τότε φάνηκε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συντονισμός ε, της ανταπόκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εμφάνιση νόσων και ανάγκη για έλεγχό τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ασθένειες και οι ιοί δεν σταματάνε στα σύνορα για να ενισχύσουμε λοιπόν τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συνεργάζεται στενά ε, με φορείς και σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον υπόλοιπο κόσμο. Για να, να σας ε, εξηγήσω τι προστιθέμενη αξία παρέχει ο οργανισμός μας. Ε, συλλέγουμε στοιχεία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι έχουμε μια συνολική ευρωπαϊκή εικόνα, μπορούμε να συγκρίνουμε δεδομένα και μοτίβα εξάπλωσης ε, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ε, σε εθνικό επίπεδο. Πριν δημιουργηθεί το σύστημα ΤΕΣΥ, ε, είχαμε διάφορα δίκτυα όπου έπρεπε τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τα στοιχεία τους. Ε, τώρα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αποτελεί μια ενιαία θηρίδη, θηρίδα, ε, εξοικονομώντας πόρους και διασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάθε μέρα στις 11.30 ε, το πρωί στο Κέντρο Πρόληψης ε, και Ελέγχου Νόσων ε, έχουμε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για να συζητήσουμε παρούσες απειλές και νέα μηνύματα που προκύπτουν στην Ευρώπη και στο υπόλοιπο του κόσμου. Με βάση αυτά, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εκπονεί μια αξιολόγηση και αξιολόγηση σχετικά με τις απαραίτητε δράσεις, αν είναι απαραίτητες. Τρίτο παράδειγμα, το Κέντρο Προλόγηση και Ελέγχου Νόσων επίσης ε, αυξάνει την ετοιμότητα των κρατών μελών ε, με προγράμματα κατάρτιση, ε, καθώς και με βελτίωση των σχεδίων ανταπόκρισης. Κατά το ξέσπασμα του ιού έμπολα, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συμμετείχε ενεργά στις δράσεις στην Γουινέα. Και πιο πρόσφατα, κατά ε, την εμφάνιση του κίτρινου πυρετού στην Αγγόλα, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συντόνισε τις δράσεις μιας ομάδας επιτόπου. Όλες οι συμβουλές και οι αξιολογήσει του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων βασίζονται στα βέλτιστα ε, διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και δεν ε, εκδίδονται με βάση εμπορικά ή πολιτικά συμφέροντα. Η ευρωπαϊκή ποικιλομορφία οδηγεί σε διαφορετικές απόψεις ε, σχετικά με τον κίνδυνο και γι' αυτό πρέπει η πολιτική, οι ε, γιατροί και η επιστημονική κοινότητα καθώς ε, και η κοινωνία των πολιτών ε, να συμμετέχουν στις δραστηριότητε μας. Ο στόχος μας είναι οι κίνδυνοι να γίνονται αντιληπτοί, να προλαμβάνονται και να ελέγχονται. Φυσικά συνεργαζόμαστε στενά με άλλους ε, οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπως ε, είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Σήμερα συνάδελφοι από την ΕΦΣΑ και το ECDC συνεργάστηκαν πάνω στην κοινή έκθεση για την μικροβιακή αντοχή που θα δημοσιευτεί εντός του έτους με τη συνεργασία μας με εμπειρογνώμονες σε όλη την Ευρώπη, ε, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εκπονεί έγκυρες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ε, πάνω σε υπάρχουσες ε, και ε, νέες νόσους. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε στο τελευταίο τμήμα της ε, ημερησίας διάταξής μας που έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων. Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της Μονίκ Γκουιάνης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Good afternoon, ladies. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέκα λεπτά έχετε. Ναι, να περιμένω να φορτώσει η παρουσίαση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προσπαθούμε εμεί πάντα να παρακινήσουμε τα θεσμικά να βελτιώσουν το πλαίσιο για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σήμερα, όπως ε, και οι άλλοι ομιλητές, βλέπω τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Πολλά από αυτά τα οποία ήθελα να πω έχουν ήδη υποθεί, οπότε θα προσπαθήσω να δώσω την πτυχή των καταναλωτών. Για να δούμε. Ε, στις γενικές παρατηρήσεις ε, θα ήθελα να τονίσω. Ε, κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι πολύ με την εμπορική πολιτική και κοιτάω τους ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες και πάντα λέω ότι ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι Ευρωπαία καταναλωτής γιατί θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το καλύτερο δίκτυο ασφαλείας στον κόσμο είτε μιλάμε για τρόφιμα, χημική ασφάλεια, κατανάλωση κτλ. Αυτό το οποίο είναι απογοητευτικό είναι ότι δεν το γνωρίζει το κοινό αυτό. Ότι αυτό οφείλεται δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν ε, το τονίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά πρέπει τα θεσμικά όργανα, οι υπηρεσίες και εμείς ε, της Κοινωνία των πολιτών να μιλήσουμε εκτός της φούσκας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα διαφορετικό αφήγημα για να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτό το δίκτυο ασφαλείας οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τα επιτεύγματα. Αυτό ισχύει βεβαίως για την ασφάλεια τροφίμων, αλλά και για άλλους τομείς ε, έχουμε πολύ ισχυρές κοινέ αρχές ε, που αποτελούν τη βάση της νομοθεσίας μας. Π.χ. η αρχή της προφύλαξης ε, όταν υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή προσέγγιση από το χωράφι στο πιάτο για την τροφική αλυσίδα. Πολύ ποιόσιμες αρχές που κάνουν το σύστημά μας τόσο καλό. Έχουμε ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο τονίστηκε ήδη και επίσης αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προς την αξία είναι η συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και συστήματα ειδοποίησης όπως το RAPEX για την ασφάλεια προϊόντων, το RASF για τρόφιμα και ζωοτροφές, κατά το οποίο κάνει το σύστημα μας πολύ καλύτερο για τους καταναλωτές και έχουμε κοινή έρευνα Ακριβώ αυτό εδώ πέρα δημιουργεί καινοτομία. Νέα α, στοιχεία τα φέρνει πολύ γρήγορα στην αγορά. Συγγνώμη, ναι. Για το περιβάλλον. Να πω το εξή. Επειδή ο Πίτερ τόνισε ε, το περιβαλλοντικό φύλλο Υπάρχει και μια πτυχή του καταναλωτή. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αυτό είναι καλό για το περιβάλλον και για τον καταναλωτή γιατί ε, θα είναι φτηνότερο να χρησιμοποιεί κανείς ε, πιο αποδοτικά προϊόντα και καλύτερο για την υγεία εάν ε, οδηγεί κάποιος σε ένα πιο καθαρό αυτοκίνητο. Το πιο καθαρό αυτοκίνητο δεν οφείλει μόνο το περιβάλλον και τη ρήπανση αλλά και σένα. Αν οδηγείς σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πιο καθαρό και εντός του αυτοκινήτου σου είσαι λιγότερο εκτεθειμένος. Πρώτα απ' όλα οι οδηγοί είναι τα πρώτα θύματα της ρήπανσης. Και επίσης, ε, κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά γνωστό, το REACH, ε, ο κανονισμός για τα χημικά. Ε, εδώ είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που έχει ο καταναλωτής δικαίωμα να γνωρίζει για τα προϊόντα, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό. Για τη δημόσια υγεία ε, τα ανέφερε ήδη ο συνάδελφος αρκετά. Αυτό το οποίο θα να τονίσω είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι όταν ταξιδεύουμε εντός της Ένωσης έχουμε πρόσβαση σε διασυνοριακή παροχή υγείας. Δεν ισχύει αυτό σε άλλα μέρη και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Μετά για την ασφάλεια των τροφίμων αναφέρθηκε. Έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα ε, ειδοποιήσεων, έχουμε ισχυρή επιστημονική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ε, με την ΕΦΣΑ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, αξιολόγηση κινδύνου. Έχουμε καλύτερους ελέγχους κινδύνου χάρη στο, ε, στο γραφείο τροφίμων και κτηνιατρικής και κάτι άλλο το οποίο ισχύει ειδικά στον τομέα των τροφίμων, ε, με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο ε, εκτεταμένη, έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε διεθνή φόρα, όπως το κόντεξ ελεμιτάριους από οποιοδήποτε μεμονωμένο κράτος μέλος. Έχει πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Αυτό ισχύει και για την ασφάλεια μου και για πολλά άλλα ζητήματα. Όπως είπαμε λοιπόν αυτή η προσέγγιση από το χωράφι στο πιάτο είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, εμποδίζει την μετάδοση των βακτηριδίων και των ασθενειών που μεταφέρονται από το τρόφιμα. Τέλος, ως τελική παρατήρηση υπάρχουν ακόμα κάποιες προκλήσεις. Η πρώτη είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για παγκόσμιες αγορές ε, και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανοίξει τους κανονισμούς της για να σταματήσουν τα λεγόμενα, οι λεγόμενοι φραγμοί στο εμπόριο. Και υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα οποία υπάρχουν ως δικλείδες ασφαλείας και στο σύστημα τροφίμων να απειλούνται από την παγκοσμιοποίηση τις ε, πολυμερεί η διμερεί εμπορικες συμφωνιες η ttip Ένωση. Είμαστε υπέρ τη παγκοσμιοποίηση των ανοιχτών αγορών, αλλά όχι τη μείωση των προδιαγραφών μας. Αυτό είναι μη ε, διαπραγματεύσιμο. Και βεβαίω, υπάρχει το κυκλικό αυτό φαινόμενο, μια, μια πίεση για απορρίθμιση και μείωση του κόστους για τη βιομηχανία, αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η ρύθμιση προωθεί την καινοτομία και έχει επίσης προλάβει σκάνδαλα και μακροπρόθεσμα. Ένα σύστημα όπου δεν χρειάζεται να έχουμε διαταραχές είναι και πιο βιώσιμο οικονομικά από ένα σύστημα στο οποίο πρέπει να παρεμβαίνουμε στο τέλος της διαδικασίας όταν έχουμε ένα σκάνδαλο. Γιατί όταν έχουμε έναν τομέα χωρίς ρύθμιση και μετά έχουμε σκάνδαλο, υπάρχει μια κοινωνικοποίηση του κόστους. Τελικά πληρώνει ο φορολογούμενος και όχι η βιομηχανία. Αυτές τις παρατηρήσεις είχα να κάνω και αναμένω βεβαίως τις ε, ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και βεβαίως ο Χίμπερτ Ντεράικε τώρα θα συνεχίσει από την ΕΦΣΑ, την Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω πέντε σημεία σε πέντε λεπτά. Ο εκτελεστικός διευθυντής ζητά συγγνώμη, είναι στην Ιαπωνία, αλλά θα έρθει την επόμενη εβδομάδα εδώ Οπότε θα έχετε ευκαιρίε να συζητήσετε αυτά τα ζητήματα. Το λέω γιατί έχουμε δύο αδελφούς οργανισμούς για να σας δείξουμε ακριβώς πόσο βαθιά είναι η συνεργασία που ανέφερε η κυρία Γκόγιας. Μια υπενθύμηση της ε, εντολής της ΕΜΣΑ. Εμείς ιδρυθήκαμε ως οργανισμός μετά από την κρίση της πογκόδους εγκεφαλοπάθειας ε, και βεβαίως ε, τις διοξίνες, αλλά αμέσως συνειδητοποιήσαμε ότι θα ήμασταν μια ρυθμιστική υπηρεσία που καλύπτει τελικά το 80% της δουλειάς μας. Επίσης θα ήθελα, δεδομένων των όσων ακούστηκαν, να τονίσω ότι η ΕΦΣΑ έχει έναν ρόλο στην ε, υγεία ζώων και φυτών και αυτό σχετίζεται με απειλές από εισαγωγές που μπορούν να καταστρέψουν το περιβάλλον μας και τη γεωργική παραγωγή. Τρία πράγματα θα ήθελα να πω για το πώς κάνουμε τη δουλειά μας. Βεβαίως θα υπάρχει κάποια επανάληψη. Το πρώτο αφορά την εμπειρογνωμοσύνη, γιατί αν δεν υπήρχαν όλοι οι ειδικοί από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις ε, δουλειέ μας. Και μιλάμε για χιλιάδες ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις που υπήρχαν και ε, όχι εκατοντάδες. Τέλος, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι δεδομένη αυτή η εμπειρογνωμοσύνη. Δεν υπάρχουν οι πόροι για να επενδύσουμε σε κάτι τέτοιο και αντιλαμβάνομαι πως οι συναδελφοί μας από την υπηρεσία φαρμάκων επενδύουν προληπτικά εδώ, κάτι το οποίο ίσως ε, δεν επιτρέπουν τα δικά μας οικονομικά. Δεν θα μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την εμπειρία στο μέλλον. Δεύτερον, σημείο συνεργασίας με τα κρατημέλη είναι ότι συνεργαζόμαστε εντατικά με τις οργανώσεις των κρατών μελών για την παρακολούθηση. Όπως ξέρετε συλλέγουμε 10 με 15 εκατομμύρια δείγματα υπολοιμάτων ζυζανιοκτώνων με διαδικασία τυποποιημένη και το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερο πάροχος τέτοιων δεδομένων. Όμως το θέμα εδώ είναι ότι Είμαστε σε επαφή με εξειδικευμένους οργανισμούς Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ολλανδία και ένα θέμα είναι ένα software που αναπτύσσουν εκεί, χρήσιμο για ολόκληρη την Ευρώπη, για μείγματα χημικών ουσιών. Αλλά το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι μια πρόκληση, γιατί χρηματοδοτούμε έρευνα υψηλού επίπεδου και πρωτογενή έρευνα, αλλά εδώ δεν μιλάμε για την καινοτόμο έρευνα, αλλά για διατήρηση συστημάτων ε, και πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα κέντρα αριστείας για να μπορούν ε, να παραμείνουν σε ηγετική θέση στο μέλλον. Τέλος, αναφέρθηκε η ΕΜΑ και η CDC και θα αναφερθεί νομίζω και η συνεργασία μας με την ΕΚΑ, αλλά πηγαίνουμε ακόμη παραπέρα γιατί έχουμε τώρα ένα δίκτυο, το EU-ANSA όπως λέγεται, οργανισμών που 13 για την ακρίβεια, που ασχολούνται με τις θετικές επιστήμες και με ζητήματα αβεβαιότητας Ελπίζουμε λοιπόν να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας με τρόπο συγκεκριμένο για να μην χρειάζεται να είστε ειδικο, ειδικοί στο κάθε θέμα και στις πτυχές της αβεβαιότητας της ε, επιστημονικής ε, εμπειρογνωμοσύνης. Έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε με το Κοινό Κέντρο Ερευνών για νέες προδιαγραφές για να έχουμε κάποια πρωτοκόλλα δοκιμών τα οποία δεν θα βασίζονται σε ζώα. Τέλος. Ε, δίνουμε, θα έλεγα, αποτελέσματα σε αρκετά χαμηλότερο κόστος από ότι αν είχαμε ε, ξεχωριστά συστήματα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε, όπως είπα, ένα σύστημα ε, μόνιμης χρηματοδότησης αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστώ. Όπως είπατε, συνεχίζουμε τον Γκέρτ Ντάνσερτ, Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών Ουσιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας εξηγήσω πώς συνεργαζόμαστε στην Ένωση για ασφαλέστερες χημικές ουσίες δηλαδή μια πανευρωπαϊκή δουλειά που γίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ουσία. Ποια είναι το αφέλη λοιπόν της συνεργασίας για τις βιομηχανικές εμπειρίες στην Ευρώπη. Ας δούμε. Καταρχάς θα έχουμε ασφαλέστερα χημικά χημικές ουσίες και χημικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα γενικότερα. Έχουμε πολίτες που θέλουν να έχουν ασφαλέστερα προϊόντα και θα έχουμε κάτι ε, we also will have efficient authorities θα έχουμε λοιπόν και αποτελεσματικές αρχές και καλύτερη χρήση των δημοσίων κονδυλίων. Η πρακτική προστιθέμενη αξία είναι ότι μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις με βάση την υψηλή ποιότητα, ταχύτητα και διαφάνεια και ανεξαρτησία και όλα αυτά νομίζω μπορούν να σας δώσουν εμπιστοσύνη στις ε, γνωμοδοτήσεις μας. Και νομίζω πως είμαστε αξιόπιστοι εταίροι των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Διαθέτοντας διάφορες πληροφορίες, συνεργαζόμενοι με πυρογνώμονες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ορίζονται από τις χώρες μέλη. Η τεχνολογία που έχουμε επίσης στην υπηρεσία μας και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους εμπειρογνώμονες και τις διάφορες εθνικές αρχές που εργάζονται πάνω στους τέσσερις κανονισμούς που διαχειριζόμαστε αποτελούν μια απόδειξη της δυνατότητάς μας να συνεργαστούμε στενά. Επίσης έχουμε και προηγμή τεχνολογία, δηλαδή λογισμικό διαθέσιμο σε επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς και εθνικές αρχές σε άλλες χώρες σχετικά με το πώς θα αποθηκεύουμε δεδομένα και πώς θα αναλύουμε τους κινδύνους των χημικών ουσιών βάσει εργαλείων που τους παρέχουμε ενημερώνοντας τα συνεχώς. Επίσης συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους. Έχουμε πάνω από 100 διαπιστευμένους οργανισμούς στην ε- Ευρώπη που συνεργάζονται στενά μαζί μας και μας παρέχουν στοιχεία όπως επίσης και την άποψή τους σε σχέση με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η υπηρεσία μας. Επίσης, προωθούν και την διαφορετική χρήση των δεδομένων, γιατί τα δεδομένα του REACH έχουν άλλη χρήση και διαφορετική χρήση από το REACH αυτό καθε αυτό. Και έτσι νομίζω βελτιώνουμε την χρήση των δεδομένων, ώστε και άλλα μέρη της Ευρώπης να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Γιατί να σας πούμε προστασία των υδάτων, ασφάλεια στο χώρο εργασία και πολλά άλλα θέματα, περιβάλλον κλπ. Επίσης, έχουμε θεσπίσει μια προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις, ενημερώνοντάς τις εκ των προτέρων για τους χημικούς παράγοντες με τους οποίους θα δουλέψουμε. Και συνεργαζόμαστε μαζί τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούν για να συλλέξουν τα στοιχεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επίσης θα πρέπει να συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας και αυτό έχει τεράστια σημασία για τις επιχειρήσεις στην Ένωση. Και με τις, επιχει... με τις χώρες μέλη μάλλον συνεργαζόμαστε όσον αφορά την ποιότητα των δομένων σε σχέση με συγκεκριμένου ε, χημικού παράγοντε, όταν υπάρχουν κάποιε ανησυχίε και αφού καθορίσουμε τι ανησυχίε, μετά χαράζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την διαχείριση αυτών των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών. Επίση, χρησιμοποιούμε τι συναντήσει μα, τι επιστημονικέ, για να κάνουμε μια επισκόπηση των επιστημονικών στοιχείων, κάτι το οποίο βοηθά και την Κομισιόν για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο δημιουργούμε μια ευρωπαϊκή αγορά συντονισμού και κοινών προσπαθειών για τη διαχείριση των χημικών και ουσιών και παραγόντων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ρωτήσω ρητορικά την προσθέμενη αξία όλων αυτών για την Ευρώπη. Θα μας το πει επόμενος ομιλητής, ο Αλεξάνδρου Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ε, να παρευρεθώ εδώ σήμερα. Θα επικεντρωθεί η παρουσίασή μου στις επιχειρήσεις και το περιβάλλον. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσω επίσης να απαντήσω σε κάποιες από τις παρατηρήσεις των προηγούμενων ομιλητών. Σχεδόν 10 χρόνια εργάζομαι στην Business Europe. Έχω συνομιλήσει με διάφορες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, μεγάλες, μικρές και μεσαίου μεγέθους. Και το πρώτο βασικό μήνυμα είναι ότι ε, η περιβαλλοντική προστασία βρίσκεται στο θεματολόγιο των επιχειρήσεων. Φυσικά μιλάμε ε, πολύ για ε, την αλλαγή του κλίματος. Αυτό όμως ισχύει και για την διαχείριση των αποβλήτων, το, την ποιότητα του νερού, την ατμοσφαιρική ρήπανση κλπ. Γιατί οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συμβαίνει αυτό. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην κοινωνία και γνωρίζουν τις ευθύνε τους. Άλλος λόγος είναι ότι είναι λογικό. Είναι συμφέρον και από ε, επιχειρηματικής πλευράς μιλάμε για την ε, καλύτερη απόδοση των ε, πρώτων υλών, των πόρων και αυτό είναι καλό και για τις εταιρείες. Επίσης έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά για παράδειγμα τις καθαρές τεχνολογίες. Ε, μια ε, αγορά που σε διεθνές επίπεδο γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Άλλος λόγος ε, είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με την νομοθεσία. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε ισχυρό περιβαλλοντικό κεκτημένο. Μπορούμε πιστεύω να είμαστε περήφανοι για αυτό το κεκτημένο και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος από το EB. Μιλήσατε για το κενό όσον αφορά την επιβολή του νόμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ξέρουμε ότι απομένουν πολλά να γίνουν όσον αφορά την επιβολή του νόμου δηλαδή εποπτεία της αγοράς και άλλα σχετικά θέματα. Ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, έχουν δεσμευτεί ε, να προστατεύσουν το περιβάλλον. Ποια είναι τα ωφέλη, ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης για την προστασία του περιβάλλοντος. Από πλευράς της βιομηχανίας ε, το πρώτο βασικό μήνυμα είναι ότι είναι σαφές ότι είναι θετική η συνεργασία. Γιατί, διότι οι επιχειρήσεις είναι ευρωπαϊκές και διεθνείς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, δρούν διασυνοριακά, αλλά και οι μικρομεσαίες συχνά έχουν πελάτες ή προμηθευτές σε όχι μόνο μία, αλλά σε διάφορες χώρες. Η ευρωπαϊκή φύση λοιπόν των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ένα θέμα κλειδί και γι' αυτό η προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος είναι λογικό να είναι ευρωπαϊκή. Θα ήθελα αυτό να σας το δείξω με διάφορα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό όμως για τη συζήτηση να έχουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα από την πλευρά της βιομηχανίας του οικονομικού τομέα. Διότι μιλάμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για την προστιθέμενη αξία που επιφέρει, που επιφέρει η Ευρώπη όταν μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικό από πλευράς του οικονομικού τομέα είναι ότι πρέπει να συγκρίνουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση με την ύπαρξη 28 διαφορετικών εθνικών καθεστώτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι το στοιχείο κλειδί στη συζήτηση. Η σύγκριση δηλαδή της ευρωπαϊκής προσέγγισης με τα 28 διαφορετικά εθνικά καθεστώτα. Η Business Europe πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση έχει αξία και έχει κυρίως ή καταρχάς να κάνει με την εκπόνηση κοινών κανόνων. Θα μπορούσα εδώ να σας δώσω διάφορα παραδείγματα όσον αφορά τα απόβλητα. Έχουμε την ε, συνεχιζόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων ε, για τα απόβλητα και τους κοινούς ορισμούς. Γίνεται πολλή δουλειά πάνω στους κοινούς ορισμούς. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία για τον ε, οικονομικό τομέα. Επίσης, ε, πρέπει να μπορούμε να συγκρίνουμε την πρόοδο που σημειώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Κατόπιν έχουμε την οδηγία για τις ε, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οδηγία αυτή αναθεωρήθηκε πριν λίγα χρόνια. Και στόχο έχει τη δημιουργία κοινών διαδικασιών κατά την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών. Έχουμε λοιπόν εδώ μια πρώτη σειρά κοινών κανόνων. Θα ήθελα επίσης να σας δώσω ένα παράδειγμα, όπως άλλωστε ανέφερε και ο κύριος Στέρν, της πιο ισχυρής φωνής που έχει η Ενωμένη Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι, πολύ, είναι απαραίτητη για να έχουμε πιο ισχυρή φωνή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Τα πιο χτυπητά παραδείγματα είναι το περιβάλλον και η, συμφωνία, η αλλαγή του κλίματος μάλλον ε, και ε, η COP21. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν καθοριστικός για την επίτευξη συμφωνίας. Ο κύριος Στέρν εξήγησε πώς πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αυτή τώρα έχουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι θα τηρηθεί η συμφωνία αυτή, κάτι που ξέρουμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα. Το τρίτο παράδειγμα που θα ήθελα να φέρω είναι η συνεργασία. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη αγορά για την ε, δημιουργία νέων τεχνολογιών και διάθεσή τους και βλέπουμε μία σειρά πλεονεκτημάτων όταν μιλάμε για την κυκλική οικονομία. Εδώ διακυβεύεται η ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς ε, πρώτων υλών. Είναι σαφές ότι όσο μεγαλύτερη η αγορά, τόσο περισσότερες οι δυνατότητες που έχουμε. Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αντί να έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα, έχουμε μία μεγάλη αγορά για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, κάτι που επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό είναι το τρίτο παράδειγμα που ήθελα να σας δώσω και το τελευταίο είναι αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος από την ΠΟΙΚ. Η συνεργασία επίσης ε, είναι, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όταν μιλάμε για την έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που σχετίζεται με τις δημόσιες αλλά και με τις ιδιωτικές επενδύσεις. 64-65% ε, των συνολικών ευρωπαϊκών δαπανών για την έρευνα και ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πολλά γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει εδώ ένα πρόσθετο επίπεδο ε, στον καθορισμό του απαραίτητου, του σωστού επίπεδου για την έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό γίνεται μέσω του προγράμματος πλαισίου Horizon 2020. Ε, αλλά έχουμε και άλλα παραδείγματα όπως είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ε, το ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν πάνω από τα εθνικά είναι απαραίτητο για προγράμματα μεγάλης εμβέλειας και είναι απαραίτητο και για τις ε, επιχειρήσεις στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι πιστεύουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στη συζήτηση όταν μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος σε εθνικό επίπεδο, μία λύση ενιαία για όλους δεν είναι πάντα η πιο κατάλληλη λύση. Γιατί? Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας για διάφορους λόγους. Έχουμε 28 κράτη-μέλη με διαφορετική ιστορία, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική γεωγραφική θέση κλπ. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να υπάρχει κάποιος βαθμός ευελιξίας. Μπορώ να σας δώσω ε, για παράδειγμα την οδηγία για τις ε, βιομηχανικές εκπομπές η οποία θέτει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, υπάρχει όμως ε, περιθώριο ευελιξίας σε τοπικό επίπεδο. Επιτρέπει δηλαδή στις τοπικές αρχές να αναθεωρήσουν ε, τα, τα όρια για τις εκπομπές. Να κλείσω λέγοντα ότι πολλά έχουν γίνει όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βιομηχανία έχει συμβάλει στι προσπάθειε ε, και συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σαφές ότι η συνεργασία, ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ενέχει πολλά πλεονεκτήματα τα οποία θα εξατμιστούν εάν επιλέξουμε να έχουμε διαφορετικά εθνικά καθεστώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάσελ Χακ, επικεφαλής της, ε, <laughs> Μονάδας. Έχετε ένα λεπτό και εγώ με δέκα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι αυτές οι πολιτικές ωφελούν όλους τους πολίτες και τους υπαλληλούς γενικής γραμματείας της Κομισιόν. Οι προλαλήσαντες ανέφεραν κάποια παραδείγματα που αποδεικνύουν την αξία που πρόσφερε η συνεργασία μεταξύ των Κομισιών και χωρών και αρχών πέραν των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα η κατάσταση είναι κάπως περίπλοκη, οπότε χρειαζόμαστε πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές πληροφορίες η παρουσία των υπηρεσιών της Ένωση σήμερα αποδεικνύει το πώς ακριβώς βοήθησε η Ένωση ακριβώς στην ε, προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Με τη χρήση ευρεία κλίμακας πόρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ήταν δυνατό αυτό. Πολύ συχνά χρειάστηκε γενικότερη δράση, γιατί μεμονωμένες χώρες μέλη ίσως δεν μπορούν να μεταφέρουν το βάρος αυτών των θεμάτων ε, χωρίς δηλαδή παγκόσμια συμφωνίες και βοήθεια. Σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε το πώς η Ένωση πραγματικά υιοθέτησε πρωτοβουλίες οι οποίες ήταν πρωτοπόρες παγκοσμίω για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Και όταν μιλάει η Ένωση, οι υπόλοιποι ακούν προσεκτικά. Παραδείγματος χάρη προστασία του περιβάλλοντος. Με ενιαία φωνή μπόρεσε η Ένωση να κάνει συμμαχίες προοδευτικές που οδήγησαν στην Συμφωνία του Παρισιού το 2015. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι τμήμα της συνθήκης, της Ένωσης, υπάρχουν κατάλληλοι στόχοι και αυτοί συνοδεύονται από απαραίτητα μέτρα που, των οποίων η εφαρμογή εποπτεύεται. Είχαμε πούμε, το σύστημα για την ε, εμπορία των ρήπων, τα συστήματα για την ε, παραγωγή χρήση γη, αλλαγή χρήση γη, δασοκομεία κλπ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν το πώ οι κοινέ προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, μέσω ανάπτυξη και παρακολουθώντα βέβαια τι μεταβολέ στην ενέργεια παγκοσμίω. Η ρήπανση βεβαίω είναι διασυνοριακή και μετά από δεκαετίες εμπειρίας έχουμε αποδείξει ότι η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική από αυτήν σε εθνικό επίπεδο για το περιβάλλον και την οικονομία. Οι παρεμβάσεις λοιπόν της Ένωσης βοηθούν την ενιαία αγορά, τις επιχειρήσεις και τις εξοικονομήσεις κλίμακος. Πράγματι, πάρα πολλές πράξεις ενιαίας αγοράς βοήθησαν εκτός από το εμπόριο και το περιβάλλον και την υγεία. Το REACH για τους χημικούς παράγοντες, η υιοθέτησή του ήταν τεράστια προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων, με στόχο την εναρμόνιση της νέας αγοράς και τη σημαντική βελτίωση του επίπεδου προστασίας σε μια πρόσφατη δημόσια διαβούλευση για το REACH, είδαμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, η βιομηχανία, η ΜΚΟ, οι οργανώσεις καταναλωτών συμφώνησαν για την προσθέμενη αξία της Ένωσης στο ΡΙΤΣ και το πώς η ε, σημασία, έχει η εναρμονισμένη προσέγγιση. Το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων στην Ένωση επιβάλλει προδιαγραφές αυστηρές και διασφαλίζει ένα προβλέψιμο νομοθετικό πλαίσιο επιτρέποντας τις επιχειρήσεις να ανθίσουν και παρομοίως οι υπηρεσίες μας διασφαλίζουν, όπως η, η υπηρεσία για τα φάρμακα, διαδραματίζουν ένα εξίσου σημαντικό ρόλο ώστε να έχουμε την βέλτιστη δυνατή προστασία υγεία των ΗΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τι Ασθένειε, για την πρόληψη και τον ελεγχό του είναι άλλο ένα εργαλείο σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε. Οι μηχανισμοί πρώιμης, πρώιμου εντοπισμού και τα μέτρα προστασίας ε, βοηθούν την αποτροπή ε, διατροφικών κρίσεων στην Ένωση ε, και προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία, εντοπίζουν τα μη ασφαλή προϊόντα και παρεμβαίνουν στην, στο εμπόριο και στις συναλλαγές ζωικών προϊόντων εντός και εκτός Ένωσης. Έχουμε πει στην εποπτεία ώστε να διασφαλίσουμε ότι για την ε, θεραπεία ας πούμε οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς ε, μορφές ε, θεραπείας. Είχαμε ας πούμε το σκάνδαλο των εφητευμάτων. που με τις δράσεις μας ανοίξαμε τον δρόμο για, νέα, για νέο ιατρικό εξοπλισμό και ο κανονισμός για, τις, τον ιατρικό εξοπλισμό in vitro υιοθετήθηκε πριν λίγες μέρες. Επίσης, ανοίγουμε, έχουμε ανοίξει και το δρόμο και για άλλες δράσεις που αφορούν τις που αφορούν διάφορες χώρες, όχι μόνο χώρες βέβαια με τις οποίες υπάρχει καθεστώς αναγνωρίσεων με την Ένωση, αλλά και άλλες χώρες όπου δεν είχαμε παρόμοιες ρυθμίσεις. Αλλά νομίζω ότι το όφελος της Ένωσης αντανακλάται ευρύτερα. Πέραν δηλαδή από την ενιαία αγορά. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Natura 2000. Είναι ένα δίκτυο 26.000 προστατευμένων φυσικών περιοχών που καλύπτει περίπου το 20% της μάζας γης της Ένωσης όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να συνεπάρξουν με ευαίσθητα και προστατευμένα ευρέως και προστατευμένους βιοτόπους. και το όφελο που προκύπτει εδώ είναι γύρω στα 200 με 300 ε, ε, δισεκατομμύρια, κάτι το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το αρχικό κόστος ε, συγκρότηση αυτού του δικτύου. Έχουμε λοιπόν εδώ την εμπλοκή όλων δημοσίων αρχών, ενδιαφερομένων, όλων ακριβώ ώστε να απολαμβάνουν όλοι από τα ωφέλη και η ανθρωπική οικονομία του Natura 2000. Παρόλο που η ρήπανση ατμοσφαιρική συνεχίζει να αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο στις πόλεις της Ευρώπης, η Ένωση πιέζει τις τοπικές αρχές, του ΣΟΤΑ γενικότερα, για την ανάπτυξη δράσεων. Είχαμε μια έκθεση περιβαλλοντική του 2015 που καταδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι σήμερα απολαμβάνουν καθαρότερο αέρα και νερού χάρη στην υψηλότερη ανακύκλωση μετά από την εφαρμογή τεσσάρων δεκαετιών νομοθεσίας. Όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύουν την προσθέμενη αξία της Ευρώπης και τέλος θεωρώ ότι και στον τομέα της δημόσιας υγείας παράγει προσθέμενη αξία η Ένωση. Παραδείγματος χάρη, η πολιτική για το κάπνισμα οδήγησε σε κάποια από τα αστρότερα μέτρα ελέγχου του καπνισμάτος παγκοσμίω. Είναι μεγάλος, είναι κύριος παράγοντας επίσης η πρωταγωνιστής μάλλον η Ένωση στο τομέα της αντιμετώπισης της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Έχουμε επίσης και τα δίκτυα αναφοράς στην Ένωση για τις ε, ασθένειες του αέρα, ώστε να έχουμε καλύτερες πιθανότητες εντοπισμού και θεραπείας. Καταλήγοντας λοιπόν, Πρόεδρε, θα θέλω να πω ότι έχουμε πολλά αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ακριβώς το πολλαπλό όφελος της Ένωσης για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των τρο... και των τροφίμων. Θα θέλαμε λοιπόν τα μηνύματα αυτά τα σημαντικά να ακουστούν και δημοσίως σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το καθήκον μας είναι να φιλτράρουμε όλα αυτά τα μηνύματα από εσάς προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα έχει φτάσει η ώρα των ερωτήσεων των συναδέλφων. Ε, πρώτα απ' όλα ο Πέτερ Λίζε, συντονιστής ε, του ΕΛΚ. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι εδώ. Νομίζω ότι το θέμα αυτό άξιζε λίγο μεγαλύτερη προσέλευση των συναδέλφων. Χαίρομαι τουλάχιστον που το ΕΛΚ είναι τα δύο τρίτα των παρόντων. Και ευχαριστώ την Μαρέιντ Μαγκίνες που είχε την ιδέα. Ε, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Τόντ Στέρν και τον κύριο Άφρε της ε, Business Europe. γιατί ε, είπε, ξεκαθάρισε το θέμα, γιατί ακριβώς είναι καλύτερη μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά σε εθνικό και ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα ναι, αρκετά πράγματα που λένε ναι, σωστά πράγματα κάνουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο. και βεβαίως ε, ε, και τελικά. Τώρα δεν είναι εδώ πέρα ε, το θέμα και ο χώρος να ζητήσετε περισσότερα λεφτά. Το θέμα μπήκε στην ημερήσια διάταξη γιατί έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Ελπίζω τέλος πάντων ε, και στη Γαλλία να έχουμε θετικό αποτέλεσμα, αλλά στο δεύτερο γύρο έχει περάσει η κυρία Λεπέν. Αν βγει η κυρία Λεπέν δεν θα μιλάμε για περισσότερα λεφτά, αλλά πώς θα εξηγήσουμε στον κόσμο τα απλά πράγματα, ότι ναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα. Ε, γι' αυτό ε, πρέπει δηλαδή να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά και παρακαλώ να τους εκπροσώπους ε, των οργανισμών. Ε, εντάξει, μιλάτε για τα τεχνικά ε, ζητήματα, αλλά και οι τρεις εκπρόσωποι των ΜΚΟ, της European Public Health Alliance και της Void, παρακαλώ να ξαναπείτε, όχι το τι θα θέλαμε, γιατί άμα τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά δεν έχει ήθελα και θα ήθελα τελείωσε. Θέλουμε ξεκάθαρα πράγματα. Τι διακυβεύεται. Αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει. Ε, δεν μιλάμε τώρα για ψηλολόγια. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει περισσότερο από ένα κράτος μέλος. Γι' αυτό ακριβώς ε, παρακαλώ να δούμε και τα καλά επιχειρήματα. Εντάξει, τα άλλα τα λέτε, να πάει στιγμή. Το θέμα μας λοιπόν είναι το μεγάλο, το χοντρό. Ναι όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πίτερ. Και τώρα ε, Μίριαμ Νταλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες τις οργανώσεις και τους εκπροσώπους των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Ε, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό. Το απλό μήνυμα ότι μαζί δηλαδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να επιτύχουμε πολύ ε, περισσότερα και η φωνή μας θα είναι δυνατότερη αν μιλάμε για την προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι μια ε, διαρκής διαδικασία. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Επιτροπή αυτή και τα μέλη της πρέπει να προωθήσουν αυτό το γεγονός σε όλες τις συνεδριάσεις, γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο σήμερα. Έχουμε συνεδριάσεις όπου μπορούμε και εμείς να εκφράσουμε στους πολίτες μας τι δουλειά που κάνουμε εδώ. Αλλά να αναφερθώ σε αυτό το οποία είπαν οι ομιλητές. Ναι, συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει μια ισχυρή φωνή όταν διαπραγματεύεται τις παγκόσμιες κλιματικές συμφωνίες και αυτό το ανέφερε η και ο κύριος Στέν και θεωρώ ότι ήταν το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η πολιτική της ε, βούληση. Και έτσι μας ακολούθησαν και άλλες περιοχές του πλανήτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο σημαντικότερος ε, σύμμαχος των ΗΠΑ με τον κύριο Στέρν, τον σύμβουλο του Ομπαμά, αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα μαζί λόγω της ενιαίας προσέγγισης που έχουμε όλα τα κράτη-μέλη. Και η Κομισιόν και ελπίζω και η Αμερικανική κυβέρνηση. Γιατί βεβαίως και η υγεία πλέον είναι ένα σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι αν είμαστε ενωμένοι ως ε, Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί ένας ομιλητής είπε ότι η υγεία είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ενδιαφέρον δεδομένων των περιορισμένων αρμοδιοτήτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. για να προωθήσουμε ακριβώς ε, τις υπηρεσίες των κατώμελών και να τις μοιραστούν μεταξύ τους και έτσι φτιάξαμε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων που είναι ένα κέντρο παγκοσμίου εμβέλειας. Και τέλος θα ήθελα να αφαιρθώ στην Business Europe που έκανα μια πάρα πολύ θετική παρέμβαση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλοί καμιά φορά θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις και το περιβάλλον δεν συμβιβάζονται. Αλλά ακούγοντα την Business Europe να λέει μεταξύ άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, βοηθάει τις επιχειρήσεις, έχουν κοινούς κανόνες, ε, ότι η συνεργασία σημαίνει μεγαλύτερες αγορές. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά και ναι, συμφωνώ ότι βεβαίως ε, η μία προσέγγιση δεν είναι ίσως η καλύτερη πάντα και ότι πρέπει να έχουμε ευελιξία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργαζόμαστε. Γιατί τελικά το ερώτημα, αν θα μπορούσαν να τα κάνουν αυτά μόνα τους τα κράτη-μέλη, αντί για μια ε, εναρμονισμένη προσέγγιση, ε, έχει μια απλή απάντηση, θεωρώ εγώ. Όχι. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω άλλο. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας και την παρουσία σας και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε τους επόμενους μήνες και χρόνια. E ευχαριστώ. Η Μαρία Μακίνες, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους ε, όσους πήραν το λόγο σήμερα το σήμερα. Όπως ανέφερε ο Πίτερ Λίζε, εγώ ήθελα πάρα πολύ ε, να γίνει αυτή η ακρόαση και θα προτιμούσα να είναι γεμάτη η αίθουσα. Φανταστείτε να μιλούσαμε για ένα σκάνδαλο, ε, για τις τιμές των τροφίμων, των φαρμάκων κλπ. Θα ήταν γεμάτη η κατάμεστη αίθουσα από ανθρώπους που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της ε, Ένωση Καταναλωτών ε, που είπε ότι χαίρεται που είναι Ευρωπαίος καταναλωτής ε, που έχουμε τόσο υψηλά πρότυπα. Δεν υπάρχει όμως ευαισθητοποίηση του κοινού. Δεν γνωρίζει το κοινό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει τόσο καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ που το είπατε δημοσίες. Σας παρακαλώ όμως να το λέτε πιο συχνά. Ε, Χθε σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Ιρλανδία είπα ότι έχουμε κάνει ζημιά στον εαυτό μας ε, τονίζοντας τα κακά αντί να σταματήσουμε για λίγο και να σκεφτούμε τι καλά πράγματα έχουμε πετύχει. διότι ε, πολλοί παράγοντε στην Ευρώπη και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις έχουν πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα και για τους καταναλωτές και για τους πολίτες μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε λοιπόν ε, αυτή την εξαιρετική παρουσίαση διότι υπάρχει ανάγκη για νέο αφήγημα και αυτή τη διαδικασία την ξεκινήσαμε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τον Πίτερ Λίζε που ε, επέτρεψε να γίνουν όλα αυτά και θα ήθελα να πω σε όλους τους ομιλητές ότι πρέπει να συνεχίσουμε το αφήγημα αυτό. Τώρα που έχω το λόγο νομίζω ότι ε, σε πολλά από αυτά τα θέματα πρέπει ε, να ακούμε τις επιχειρήσεις, τους πολίτες μας, μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και επειδή συνεχίζεται και η συζήτηση για το Brexit, θα πρέπει να ακούσουμε αυτούς που φοβούνται ότι θα χάσει και η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποσυρθεί τελείως από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Κάτι που ελπίζουμε να μην γίνει και λόγω της ε, συμβολής του στην ε, έρευνα και καινοτομία. Αλλά ε, άλλο σημαντικό ερώτημα είναι στην πράξη απόσυρσης που θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό το Ηνωμένο Βασίλειο. Μου φαίνεται ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να συνεχίσει να συμμετέχει στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διατηρηθούν τα πρότυπα που εφαρμόζει και το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή. Οι εμπειρογνώμονε μας εδώ σήμερα έχουν σκεφτεί το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας. Ναι, πολύ σωστά. Και ελπίζω οι εμπειρογνώμονες μας να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Η Κάριν Κάντεμπαχ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω θερμά την Μέιραντ Μακίνε για την πρωτοβουλία αυτή, διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Το κοινό έχει την εντύπωση ότι η πολιτική είναι απλά ο αγώνας για επικράτηση μιας θέσης. Το ότι όμως έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα, συχνά ξεχνιέται. Έκκλησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επικοινωνιακή στρατηγική της ε, να κάνει περισσότερα. Ακούσαμε ότι υπάρχουν ε, πολλές καλές υποθέσεις που θα πρέπει να ακουστούν ε, και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να τονίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει σε διάφορους τομείς. Στις συζητήσεις με τους ψηφοφόρους μας ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μεταφέρουμε όχι μόνο αυτά που δεν έχουμε πετύχει, αλλά και αυτά που πετυχαίνουμε στην ε, καθημερινή δουλειά μας ε, στον τομέα της υγείας ε, και σε πολλούς άλλους τομείς. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι κάτι που ξεχνιέται τελείως. Και είναι κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε όχι μόνο στο πλαίσιο των επομένων εκλογών. Και Πέτερ Λίζε, συχνά συμφωνώ με τις θέσεις σου, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι αιτιολογημένο το αίτημα για περισσότερους οικονομικούς πόρους. Όταν επιβάλλουμε νέες υποχρεώσεις στους οργανισμούς μας θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να έχουν και την αντίστοιχη χρηματοδότηση. διότι αλλιώς ε, δεν μπορούν ε, να εκπληρώσουν τις ε, υποχρεώσεις τους οι οργανισμοί αυτοί. Και μιλώ ως εισηγήτρια του θέματος των επίσημων ελέγχων. Όταν λοιπόν περιμένουμε η ΕΦΣΑ ή το Κοινό Κέντρο Ερευνών να πληρεί τις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να έχουν και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Διότι αλλιώς θα λάβουμε εκ των υστέρων το λογαριασμό. Δηλαδή μας επιβάλλατε ένα σωρό υποχρεώσεις, ένα σωρό καθήκοντα, αλλά δεν είχαμε τα απαραίτητα μέσα για να το πετύχουμε. Σε μια τέτοια συζήτηση, λοιπόν, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η συζήτηση για τους απαραίτητους πόρους. Ελπίζω τη συζήτηση που είχαμε σήμερα να μπορέσουμε να την έχουμε πιο συχνά στο μέλλον. Νομίζω ότι έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα και όσο περισσότερο τα συζητάμε, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνουν και αντιληπτά. Πρέπει να επαναλάβει κανείς κάτι πολλές φορές προτού γίνει κατανοητό. Έχουμε λοιπόν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να τη μεταφέρουμε στους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σέικχαουτ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέρφους μου που ε, ανέφεραν το πόσο επήγει αυτό στη συζήτηση. Ακούσαμε πολλά, αλλά τελικά το θέμα είναι τι διακυβεύεται μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ με σένα Λίσε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπερασπιστούμε αυτά που έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ. Αλλά πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τις τάσεις στις κοινωνίες μας όπου μειώνεται η υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τι μπορεί να κάνει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην μειωθεί περαιτέρω η υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ας είμαστε ειλικρινείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται ε, οντότητα που προστατεύει όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα όχι ε, τους λιγότερο μορφωμένους που πιστεύουν ότι χάνουν στην, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης Κοιτάξτε τις ε, εκλογές ε, στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, παντού. Ε, συνήθως το μισό του πληθυσμού είναι εναντίον, που θεωρούν ότι δεν ότι δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντά του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει, μόνο, στην Ευρώπη και χαίρομαι πολύ που είναι ο Τότ Στέρν εδώ πέρα. Ε, η ερώτησή μου λοιπόν απευθύνεται στον Αλεξάνδρ Άφρε από την Business Europe. Εντός της Business Europe πραγματοποιείται συζήτηση με καινοτόμα προσέγγιση ε, διότι η αλλαγή της συνθήκης είναι ταμπού εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Βρυξελών. Αλλά θα ήλπιζα η Business Europe να σκέφτεται με πιο καινοτόμο τρόπο. Το παρόν θεσμικό πλαίσιο βλέπουμε ότι εποφελούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι επιχειρήσεις. Έχουμε την εσωτερική αγορά, ε, ε, έχουμε αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά έχουμε και φορολογικό ανταγωνισμό, διότι δεν θεωρείται η φορολογία ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι και εμείς θα από τον φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά αυτό μειώνει τα έσοδα των κρατών μελών, ε, δηλαδή λιγότερους πόρους για την κοινωνική ασφάλιση, για παράδειγμα, και μαντέψτε ει βάρο ποιου γίνεται αυτού, αυτών που ούτω ή άλλω χάνουν από την παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική, τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πετύχουμε σε αυτόν τον τομέα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ θα ήλπιζα η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, βελτιωθεί μόνο στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλε τι πτυχέ ε, και αυτή είναι η ερώτησή μου προς τον Πέτερ Να ευχαριστήσω τον Τότ που βρίσκεται εδώ. Ήταν η πρώτη σας δημόσια ομιλία σήμερα, αλλά έχουμε συναντηθεί κατηδίαν επανειλημμένα. Ε, όλοι νομίζω θα ήθελαν να ακούσουν τη θέση σας ε, σχετικά με το εξής. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει η απόσυρση του σχεδίου για την καθαρή ενέργεια ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι συμβολική η κίνηση αυτή ή πιστεύετε ότι θα δούμε σημαντικές αλλαγές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τελευταία ερώτηση. Ήδη αναφέρατε πόσο σημαντικό θα είναι το θέμα αυτό για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ε, ξέρουμε όμως ότι το 2018 οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν θα μας δώσουν αυτά που περιμένουμε. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι δεσμεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, δεν θα αρκέσουν ε, ούτε για συγκράτηση κατά 2 βαθμούς Κελσίου, ούτε κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Τι θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε το 2018 για να έχουμε περισσότερη φιλοδοξία και δεν θα πρέπει να παίξει και εδώ κάποιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη του πολύ έμπειρου Τότ Στέρνς. Uh, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιούσο, ο τελευταίος ομιλητής. Μετά από αυτήν κλείνει ο κατάλογος και θα ζητήσω από τους καλεσμένους μας να απαντήσουν. Κυρία Γιούσο, ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των υπηρεσιών που ήταν σήμερα εδώ και τους οργανωτές αυτής της ακρόασης. Οι υπηρεσίε νομίζω δίνουν προσθέμενη αξία την οποία αγνοούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει να τη διαφημίσουμε περισσότερο και να δείξουμε τις συνεργασίες μας και το πόσο καλές είναι για την Ένωση. Και επιτρέψτε μου να κάνω συγκεκριμένο ερώτημα στο Διευθυντή της Υπηρεσίας για το Περιβάλλον γιατί αναφέρθηκε στα 20 μιλιγράμμ καδμίου ένα κιλό. Να ρωτήσω αν έκαναν μελέτη ή αξιολόγηση κινδύνου επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τοξικότητας συστήνει να γίνει μια αξιολόγηση κινδύνου πριν τον καθορισμό των όριων. Το Νοέμβριο του 2015 η ίδια Επιτροπή είπε ότι κάτω από τα 80 μιλιγκράμμ ανά δεν υπάρχει συσσόρευση καθημερινή στο έδαφος. Η Κομισιόν έλαβε ως αναφορά την νομοθεσία σε χώρες όπως η Σουηδία όπου η γεωρική δραστηριότητα είναι χαμηλή και ο φωσφορίτης περιέχει ελάχιστο κάδμιο. Όμως στις χώρες του Νότου με υψηλή γεωργία και με φωσφορίτη από άλλες περιοχές δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και η αποκαδμιοποίηση σήμερα είναι στην ουσία αδύνατη βιομηχανικά. Να ρωτήσω λοιπόν, μήπως έχετε κάποια μελέτη σε σχέση με τη σύσταση αυτή. Μετά, για την έλλειψη πόρων, για την ΕΣΑ που πραγματικά κάνει πολλή δουλειά και έχει πολύ φόρτο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι δεν συλλέγει φόρους, αλλά άλλοι συλλέγουν φόρους υπέρ μεγαλύτερης ανεξαρτησίας Οπότε θα έλεγα δεν ξέρω τι γίνεται με την επιβολή φόρων ή όχι, γιατί υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που επιβάλλουν φόρους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή όχι. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν το Business Europe, οπότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το Business Europe. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν υπήρξαν τόσε ερωτήσει άμεσα για μα. Σχόλια είχαμε για το Business Europe. Πάντως, να αναφερθώ σε τρία σημεία, αν θέλετε. Πρώτον, από τα σχόλια διαφαίνεται η ανάγκη περισσότερης προβολής για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Εδώ ακριβώς λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες έχουν ένα σημαντικό ρόλο μέσω των δραστηριοτήτων τους. Και εγώ κρατάω τις προτάσεις που άκουσαν επαγγελμένως γι' αυτό. Αυτή είναι η πρώτη μου τοποθέτηση. Η δεύτερη αφορά κάτι που είπε η κυρία Μαγκίνες Γκρέν, ήταν ερώτηση για το ETS ε Εδώ με το Brexit δεν μπορώ να απαντήσω πλήρως. Δηλαδή, βέβαια, ό,τι και να γίνει βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, δεν θα πρέπει να υπάρχει βλαβερή επίπτωση στο ευρωπαϊκό ΙΤΕΣ που άλλαξε στην Ευρώπη. Και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Πάντως από ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα, ο αντίκτυπος θα αφορά το ETS ε, της Ένωσης και θα είναι σχετικά χαμηλό. Χαμηλός ο αντίκτυπος. Μετά. Μια άλλη ερώτηση χάσει νομίζω. Προσπαθούμε, δεν είναι πάντοτε εύκολο στις Βρυξέλλες, αλλά συνεχίζουμε τις προσπαθίες μας. Δεν θα σχολιάσω βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι εγώ αρμόδιος ας πούμε για θέματα όπως η φορολόγηση. Και στο συγγνώμη, αλλά ελπίζουμε να μην, να μην μάλλον αποκομίσατε αυτό από τα σχολιά μου όταν μιλούσα για προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, να μην μείνουμε μόνο στην τωρινή κατάσταση στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι τα πράγματα θα πρέπει να προχωρήσουν, θα πρέπει να υπάρξουν αναθεωρήσεις, αξιολογήσεις, πρόοδοι, ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά. Και, και εμείς θα συμμετάσχουμε στο, στη συζήτηση για το πολυδιάστατο μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχουν πτυχές περιβάλλον, υπάρχουν πτυχές ενέργειας, οπότε οπωσδήποτε θα συμμετάσχουμε και εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε επειδή υπήρξε μια ερωτήσει και για εσά παρακαλώ. Και εγώ βεβαίω, θα τα ξαναδώ αυτά. Το διοικητικό μα συμβούλιο αποφάσισε ότι και εμεί πρέπει να συνεισφέρουμε σε ένα καλύτερο αφήγημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την άμεση ερώτηση του κυρίου Λίζε. Θεωρώ ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ενιαία αγορά, είναι μια αγορά. Αν επανεθνικοποιήσουμε ε, τα πράγματα αυτά πηγαίνουμε στην αντίθετη κατεύθυνση του πού πηγαίνουν οι αγορές. Ε, είναι παγκόσμιες εταιρείε, παγκόσμιες αγορές, ψηφιακές αγορές. Οπότε, εάν ε, δώσουμε την αρμοδιότητα εποπτείας και ρύθμιση αυτών αγορών στις χώρες, μετά ξεκινάει μια περιδίνηση γιατί μετά θα έχουμε αρνητικό ανταγωνισμό για τους ε, κανόνες, ε, λίγο ανταγωνισμό μεταξύ των εθνικών αρχών, θα χαθεί το δίκτυο ασφαλείας για τους καταναλωτές και μια λιγότερο αξιόπιστη αγορά. Γιατί δεν θα έχουμε μετά και ίσους όρους ανταγωνισμού κτλ. Οπότε ε, είναι ένα σενάριο το οποίο πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία γιατί η Ευρώπη μας έχει φέρει ένα επίπεδο αξιοπιστίας και ασφάλειας ε, πολύ καλό. Και βεβαίω πάντα θέλουμε περισσότερο, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση, αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να αποδομήσουμε αυτό το οποίο χρειάστηκε δεκαετίες για να οικοδομηθεί. Να πω και κάτι για τον Brexit. Γιατί οργανώνουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο μια διάσκεψη για τον Brexit και τα θετικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές αλλά οπωσδήποτε αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το ότι οι καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου κινδυνεύουν να μην καλύπτονται από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να σημαίνει κάποιες ευκαιρίες στους τομείς όπου θα είναι πιο φιλική η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά σε άλλους τομείς θα χάσουν ένα σύστημα προστασίας επειδή δεν θα είναι πλέον πολίτες της Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά θα χάσουν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν αυτό ερώτημα. Υπήρχε ένα ερώτημα και προς τον καλεσμένο μας από τις ΕΙΠΑ. Χαίρομαι πάντα να ακούω ερωτήσεις από τον φίλο μου τον Μπάς Άικχαουτ και θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση για την καθαρή ενέργεια και το εάν ε, η ανάκληση του σχετικού νόμου είναι συμβολική ή αν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, νομίζω πως είναι ένα μείγμα προόδου προς τον στόχο του 32% μείωση των εκπομπών στον τομέα της ενέργειας μέχρι το 2030 που έχουμε προχωρήσει ήδη αρκετά ε, στην πράξη και όμως νομίζω ότι το σχέδιο αυτό καθαρής ενέργειας ε, και το πώς ε, διαμορφώθηκε είχε στόχο να προωθεί στην ανανεώσιμη ενέργεια, την αποτελεσματική χρήση και νομίζω ότι θα δούμε πια λιγότερα τέτοια πράγματα Το άλλο το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν εστιάζει μόνο εκεί, αλλά στόχο έχουν να μειώσουν κάποια από τη φιλοδοξία που υπάρχει στις προδιαγραφές ε, οχημάτων, όπου πηγαίναμε από τα 27 στα 44 μίλια να η κατανάλωση σε μια περίοδο 12 ετών και θα το επανεξετάσουν αυτό. και θα έλεγα ότι υποβαθμίζονται οι κανονισμοί που έγιναν επί Ομπάμα για το μεθάνιο για διάφορους τομείς. Είναι μια ευρύτερη προσπάθεια πέρα από τα εργοστάσια ενέργειας όσον αφορά... Γενικά νομίζω ότι θα υπάρχει απτός αρνητικός αντίκτυπος ε, των πολιτικών ε, Τραμπ. Ε, Α, εντάξει, θα είναι πλήρης αναστροφή ή κάτι τέτοιο. Τώρα, για το πώς θα διατηρηθεί η φιλοδοξία θεωρώ ότι είναι σημαντικό, αν θα έρθει η φιλοδοξία, είναι σημαντικό στο πλαίσιο του να εστιάζουμε στην ανάπτυξη και την ισχύ του συστήματος των Παρισίων να μην ε, χάνουμε να μην ξεχνάμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα αναπτυχθούν ε, στα συστήματα τα σχετικά με το Παρίσι, κατευθυντήριες γραμμές ε, και διαφόρων ειδών κατευθύνσεις ε, που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευση για να τελειώσουμε το 2018 και το σημαντικότερο νομίζω αφορά την διαφάνεια και κάποια ζητήματα χρηματοδότησης. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, δηλαδή αν γίνουν λάθος, αν γίνουν με έναν τρόπο ε, ουσιαστικό νομίζω θα έχουν κάποιο σημαντικό αντίκτυπο για την φιλοδοξία την ίδια θα έλεγα το που θα πάνε οι στόχοι θα έχουμε μια αρχική θα έλεγα εξέταση του τι θα κάνουν οι χώρες στο σύνολό τους το 2028 και το 2020 είναι το σημείο στο οποίο θα δούμε τους ε, συγκεκριμένους στόχους και ελπίζω να αυξηθούν. Τέλος, όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο είπα δεν συμμετέχουν σοβαρά στις διαπραγματεύσεις, αυτό Μυρία, θα έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο. Αυτό το οποίο θα δούμε νομίζω στις ΗΠΑ είναι το ότι υπάρχει ήδη στο υποεθνικό επίπεδο σοβαρή δράση, δηλαδή κάποιες πολιτείες και πόλεις νομίζω μία περίοδο συγκρίσιμη από το 2001 με το 2008 που θα έλεγα ότι οι είχαν ε, βρεθεί στο περιθώριο όσον αφορά την ε, κλιματική αλλαγή. Υπάρχει κοινωνία των πολιτών, εταιρείε κτλ. Στην πραγματική οικονομία δηλαδή όσον αφορά την καθαρή ενέργεια. Αυτό θα συνεχιστεί αλλά είπα, ως κινητήριος δύναμη δεν νομίζω να συνεχίσει να έχει τον ίδιο ρόλο. Και προφανώς έτσι η συνεισφορά της Ένωσης είναι ακόμη σημαντικότερη. Το άλλο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι το εάν θα παραμείνουν στη συμφωνία του Παρισιού ή όχι. και θα έλεγα εντάξει είμαι συγκρατημένα ε, αισιόδοξο ε, ότι σε τελική ανάλυση η κυβέρνηση θα παραμείνει εντός της συμφωνίας ίσως θα προτείνουν κάποιες αλλαγές Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εντός της κυβέρνησης ε, και μεγάλες εταιρείες και οι εταιρείες ε, ορυκτών καυσίμων είναι υπέρ τη συμφωνία ε, του Παρισιού. Και βεβαίω παίζουν ένα ηγετικό ρόλο και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή αλλά και τις παράπλευρες απώλειες που θα υποστούν οι ΙΠΑ εάν φύγουμε. Εγώ νομίζω ότι θα παραμείνουμε συμφωνία αλλά είναι ανοιχτό θέμα. Μάλιστα θα δούμε τι θα συμβεί. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς μας γιατί με ενημέρωσαν ότι πρέπει να τελειώσουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, Πέντε λεπτά στα αγγλικά. Βεβαίω είδα τον Πίτερ και την Νίνα. Θα σας δώσω τον λόγο για να δώσετε απαντήσεις. On, on that, I, I don't know who to choose. As I would say, any, mini, mini, mo. Geert, do you think you could, you can, you, you could try to answer? Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το βασικό στοιχείο που προκύπτει από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι γνωστό στους πολίτες μας ε, τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες από την πλευρά μας να βελτιώσουμε την επικοινωνία όσο μπορούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό στοιχείο και σημαντικό είναι να μην σταματήσουμε να καταβάλουμε τις προσπάθειες αυτές. Ο τύπος γενικά δεν ενδιαφέρεται για τα καλά νέα. Νομίζω ότι οι δραστηριότητες μας αναφέρονται πολύ στον εξειδικευμένο τύπο. και επίσης οι καταναλωτές που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτικών μας επίσης ενδιαφέρονται. Και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δηλαδή ενδιαφέρονται. Αλλά νομίζω ότι για να ενδιαφερθεί περισσότερο ο γενικός τύπος ε, θα πρέπει να καταβληθούν ε, προσπάθειες από τις Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι νομίζω ε, έχουν ε, καλύτερες δυνατότητες να κινήσουν τα πράγματα στον γενικό τύπο. Επίσης, όσον αφορά τις ε, περικοπές ε, των πόρων και ιδιαίτερα μετά το Brexit και την δυνατότητα ίσπραξης τελών. Θα επικροτούσα οι οργανισμοί να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κατά την παροχή υπηρεσιών ε, σε επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη, εισπράττοντας τέλη, ώστε να, είναι πιο, ώστε να μην επηρεάζονται τόσο πολύ από περικοπές στη χρηματοδότηση, για να μπορέσουμε καλύτερα να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω ότι αυτό θα το επικροτούσαμε και ελπίζω στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ανοιχτή απέναντι σε τέτοιες λύσεις που πιθανότατα να απαιτούν τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν προς όφελος όχι μόνο των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με το